Καλησπέρα σας. Συμπαθάτε που αρχίσαμε ε, με καθυστέρηση. Αλλά να βλέπετε, φοράω την Ιρλανδική Πράσινη Προεδρία. Ε, γι' αυτό άργησα, με κάλεσε η Ιρλανδική Προεδρία και ήταν εκεί όλοι ε, εκεί πέρα, 27, 27 εκπρόσωποι από τα κρατημέλη και έγινε μια συζήτηση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Βέβαια και ο Χάνης θα σας το επιβεβαιώσει. Ο καλός μας φίλος, ο κύριος Σεμέτα, είναι αδιάθετο σήμερα, ήθελε πάρα πολύ να έρθει. Και ε, θα έπρεπε να σηκωθεί από το κρεβάτι του πόνου εδώ, αλλά ο Χάιν Σούρεκ, ε, ο οποίος ε, είναι παλιό γνωστό από την Γενική Διεύθυνση τη επιχειρήση. Ήρθε αντί του κύριου Σεμέτα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθε να μας Και συζητήσαμε ακριβώ αυτά που είχε να μας παρουσιάσει και είπαμε ε, μεθοδολογικά να σας προτείνουμε το εξή. Πρώτα πρώτα θα μα μιλήσει για τον τελωνιακό κώδικα, τον ενιαίο τελωνιακό κώδικα θα γίνουν ερωταπαντήσεις και στη συνέχεια θα μας μιλήσει για τα γενικότερα ζητήματα τα οποία μας ενδιαφέρουν. Και ας μην είναι μερικά από αυτά ε, στις στενή ενία e e αρμοδιότητες μας. Εάν συμφωνείς, πρέπει να φύγεις. Στη τρεις ώρα κάποιος άλλος θα έρθει. I'm on British time. <laughs> um, four o'clock. στις τέσσερις, στις τέσσερις. Thank you very much for... Σας ευχαριστώ που με καλέσατε και μου τηλεφώνησαν σήμερα το πρωί να πήγαινα στο αεροδρόμιο και μου ζήτησε ο Επίτροπος να τον αντικαταστήσω. Ήταν να φύγω για το Βερολίνο, όπου θα συζητούσαμε το θέματα ε, της ε, φοροδιαφυγής στην Bundestag. Να λοιπόν, ε, πώς ε, υπάρχει ένας σίγουρος τρόπος για να εξελίσσεται έσοδα και το κράτος μέσω των τελωνίων. Με μεγάλη μου χαρά σας ξαναβλέπω. Γιατί επίση θα πρέπει να σας πω πόσο σας είμαι ευγνώμων διότι η Επιτροπή σας έχει πάρα πολύ υπεύθυνη, σοβαρή στάση όσον αφορά την προβληματική για τον ελληνικό κώδικα. Και θα πρέπει να παραδεχθώ ότι και στο Συμβούλιο είμαστε αποφασισμένοι ούτως ώστε η υπόθεση αυτή να προωθηθεί. Πάντως, εάν με επιτρέπετε, να σας πω πάρα πολύ σύντομα για ποιο πράγμα θα συζητήσουμε. Γιατί μετά θα αρχίσουμε τα πιο τεχνικά θέματα, θέματα τακτικής. Να, έχω ένα σύντομο βίντεο το οποίο έχουν προετοιμάσει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 Νομίζω ότι ήταν σύντομο, αλλά νομίζω ότι καταλάβατε πόσο σημαντική είναι η Τελωνιακή Ένωση ε, και πόσο μεγάλη σημασία έχει για την ζωή των πολιτών της Ευρώπης. Αυτό που θα κάνω σήμερα είναι ότι θα ασχοληθώ με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως είπε και ο Μάλκον. Θα ξεκινήσω με τον <coughs> εξυγχρονισμό της νομοθεσίας για τα τελωνία και να σας πω ποιες είναι οι άμεσες προτεραιότητες. Uh, και μετά θα αναφερθώ στους προσανατολισμούς ε, τους γενικούς αλλά και σε κάποια θέματα ΦΠΑ που ενδεχομένως δεν είναι άμεσα ε, του δικού σας ε, πεδίου αλλά παρόλα αυτά πρέπει να το αναφέρω. Για μία ακόμα φορά να σας ευχαριστήσω όλους και εσάς προσωπικά και όσους ε, δουλεύουν για τον τελωνιακό κώδικα. Να τους ευχαριστήσω, λέω, για την εξαιρετικά επικοδομητική του στάση και την αφοσίωση με την οποία ασχολούνται με το ε, θέμα αυτό. Πρέπει να μην λησμονούμε ότι αυτό το οποίο κάνουμε εμείς εδώ είναι στην ουσία να καθορίζουμε τους κανόνες για όλες τις τελωνιακές αρχές των 27 χωρών που σύντομα θα γίνουν άλλωστε και 28 έτσι ώστε όσο γίνεται πιο αρμονικά και εναρμονισμένα να εφαρμοστούν οι ίδιες ε, αρχές έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τα ίδια δεκυβεύματα, οι ίδιες προκλήσεις με όσο γίνεται πιο ομοιόμορφο τρόπο. Και επίσης να μην λησμονούμε ότι με τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε στην καλή λειτουργία και της εσωτερικής αγοράς αλλά και του εξωτερικού εμπορίου. Πάντα έχοντας σαν κύριο γνώμονα πλέον την ασφάλεια των πολιτών ε, και καταναλωτών μας. Δεν είναι μια κίνηση ξαφνική. Ξεκινήσαμε το 2003 προσπαθώντας να εξυγχρονίσουμε ε, τους ε, κανόνες των τελωνίων. Γιατί μη ότι η ολοκλήρωση των τελωνίων ήταν ένα από τα πρώτα και πιο σημαντικά βήματα που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν ε, ένα από τα μεγαλύτερα βήματα αυτή η Τελωνιακή Ένωση της σύγχρονης Ευρώπης. Τα τελευταία χρόνια ε, προσπαθήσαμε να κάνουμε μια εξωτερική ε, αξιολόγηση που βασίζεται και στους εξωτερικούς ε, operators, ε, στους εξωτερικούς ε, εμπλεκόμενους φορείς και άλλους που ασχολούνται με το θέμα. Και επομένως θέλουμε να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα τα οποία δεν θα ε, βοηθούν έτσι ώστε να αναπτερωθεί το δικό μας ε, ηθικό ή ε, ο εγωισμός μας, να πούμε τι ωραία τα κάνουμε όλα, αλλά να δούμε πώς μας βλέπουν και πώς μας αξιολογούν οι εξωτερικοί μας εταίροι. Σας ορκίζομαι ότι η Κομισιόν παρακολουθεί όλο αυτό το σήμα, το σχέδιο συγγνώμη, και το θέμα από πάρα πολύ κοντά ε, και ο Επίτροπος ε, ε, Σεμέτα ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το θέμα και μάλιστα βιαζόμαστε γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Είμαστε πιεσμένοι. Πρέπει να γίνει η αναθεώρηση πριν τεθεί σε ισχύ το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. και θα πρέπει λοιπόν η αναθεωρημένη Τελωνιακή Ένωση να αρχίσει να ισχύει, να ισχύει άμεσα. Έλαβα την ε, έκθεση με, το, με την έκβαση του χθεσινοβραδινού, χθεσινοβραδινού τριμερούς ε, διαλόγου. Φαίνεται να ε, έχει πάει καλά. Και βεβαίως υπάρχει και ένα άλλο που θέλω να σας πω είναι ότι δουλέψατε όλοι πολύ στενά και σε στενή συνεργασία με την ε, Προεδρία όσον αφορά, τις, ε, όσον αφορά την ε, ενδυνάμωση και την εφαρμογή, την υλοποίηση των αποφάσεων, γιατί ε, αυτή τη στιγμή προχωρήσαμε και λίγο σε αχαρτογράφητα ύδατα. Μετά από την ε, συνθήκη της Λισαβόνας ξεκινήσαμε σε περιοχές τις οποίες δεν γνωρίζαμε πολύ καλά. Είμαστε αισιόδοξοι, πολύ αισιόδοξοι, ότι στον επόμενο γύρο του διαλόγου τον Απρίλιο θα καταφέρουμε να επιτύχουμε συμφωνία μεταξύ των διοθεσμικών οργάνων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα του διαλόγου. Ε, το βέβαιο είναι ότι σε πνεύμα συνεργασίας οι δύο συνομοθέτες μπορούν να προχωρήσουν καλύτερα. Έχουμε δουλέψει πολύ σκληρά και αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι εξίσου σημαντικό να έχουμε και αποτελέσματα. Ε, και ε, ε, βεβαίω πρέπει να σας πω ότι οι εμπειρογνώμονε μας είναι πάντα στη διάθεσή σας έτσι ώστε να σα δώσουν οποιαδήποτε τεχνική αρρωγή θα χρειαστείτε οποιαδήποτε στιγμή. Δύο λόγια για το χρονοδιάγραμμα. Δηλαδή αν θα τα καταφέρουμε έγκαιρα να ολοκληρώσουμε την εργασία. Σχετικά με αυτό και ε, το Συμβούλιο και ο Επίτροπος έχουν αυτό στο νου τους. Και πρέπει να σας καθησυχάσω ότι δηλαδή δεν θα υπάρξει κανένα νομικό κενό στον τομέα αυτό έστω και αν όταν συμφωνήσουμε επί της ουσίας τον Απρίλιο είναι ε, πλέον πολύ αργά έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Τούτη τη στιγμή στην Κομισιόν ε, προσπαθούμε να βρούμε μία ενδιάμεση λύση έτσι ώστε οποιαδήποτε στιγμή, έστω και για μία ώρα, να ε, μην υπάρξει νομικό κενό. Θα προκύψει κάτι λοιπόν το οποίο θα μας δώσει αρκετό χρόνο έτσι ώστε να ολοκληρώσουμε ορθώς την ε, διαδικασία. Και είναι κάτι ε, το οποίο έχουμε συζητήσει μαζί σας και βεβαίως έχουμε ακούσει τις ανησυχίες σας όπως έχουμε ακούσει και τις ανησυχίες των εμπορευομένων. Σας υποσχόμαστε λοιπόν εξ αρχής ότι μέχρι τον επόμενο τριμερή διάλογο θα έχουμε απάντηση σε αυτό το κέριο ερώτημα, δηλαδή ε, πώς θα βρεθεί αυτή, ε, αυτό το plan B ε, και πώς θα υλοποιηθεί αυτό το plan B έτσι ώστε να μην υπάρξει νομικό κενό. Αυτό όμως δεν πρέπει να μας ε, ε, ε, από, να, να, να στρέψει την προσοχή μας από το συγκεκριμένο ζήτημα που μας απασχολεί και που πρέπει να είναι και ο τελικός μας στόχος. και νομίζω ότι ε, είναι η στιγμή τώρα που ανάλογα με τις κινήσεις που θα πάρουμε θα σταματήσουμε να είμαστε πειραματόζωα και θα είμαστε πλέον σκαπανείς και πρωτοπόροι. Έχουμε πολλά πράγματα στα σκαριά. Και στόχο αυτό τα έχουν μεταξύ άλλων τη σωστή υλοποίηση των διανοητικών δικαιωμάτων. Η οδηγία θα είναι πολύ σύντομα έτοιμη και σίγουρα πολύ γρήγορα θα έχουμε και τις εκτελεστικές πράξεις οι οποίες πρέπει να την συνοδεύουν έτσι ώστε να ε, υπάρχει ε, η ε, άμεση πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται έτσι ώστε να υπάρξει άμεση δυνατότητα κατάσχεσης ας πούμε, άμεση πρόσβαση στο προϊόν και άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες των τελωνίων, συγγνώμη, άμεση πρόσβαση των τελωνίων στις πληροφορίες πληροφορίες ε, για ε, παραχαραγμένα προϊόντα. Επίσης, Έχουμε και το νέο ε, σχέδιο δράσης των τελωνίων για τις διαδικασίες παραβίασης των διανοητικών δικαιωμάτων. Έχουμε προετοιμάσει ήδη ε, και το, τα ε, ζητήματα τα οποία αφορούν και την εποπτεία της αγοράς αλλά και την ε, προστασία των προϊόντων. Όσον αφορά την εποπτεία της αγοράς πρέπει να σας πω ότι είχα αρχίσει να ασχολούμαι ήδη με το θέμα αυτό στη Γενική Διεύθυνση Enterprise και τώρα βλέπω το ίδιο θέμα από άλλη πλευρά η εποπτεία της αγοράς έχει ένα ευρύ φάσμα ο τελωνιακός κώδικας μαζί με την εποπτεία της αγοράς πρέπει να δώσει την δυνατότητα στους υπευθύνους των τελωνίων να ελέγχουν γρήγορα και αποτελεσματικά όλα τα εισαγόμενα ε, αγαθά και προϊόντα πρέπει να κινηθούμε με τρόπο ε, ενεργητικό έτσι ώστε να ξεπεράσουμε τα υφιστάμενα προβλήματα. Σε αυτό ξέρω ότι μπορούμε να ε, υπολογίζουμε και τη δική σας βοήθεια και το δικό σας, ε, τη δική σας στήριξη. Έχουμε λοιπόν και την προσέγγιση των εθνικών ε, καθεστώτων για την, στα πλαίσια του νέου κώδικα, γιατί Ξέρετε, ε, ε, υπάρχουν διαφορές, δηλαδή μία παράβαση ε, μπορεί να είναι εγκληματική παράληψη σε μία χώρα, απλή παράληψη που επισύρει κάποιες κυρώσεις σε άλλη και πράξη για την οποία ο υπεύθυνος θα λάβει μια απλή παρατήρηση ή προειδοποίηση, ας πούμε. Ο βαθμός των κυρώσεων διαφέρει από χώρα σε χώρα, όμως χρειάζεται ομοιογένεια και των κυρώσεων, ε, δηλαδή η ε, συμπεριφορά, οι κανόνες και οι κυρώσεις μετά από ε, παραβατικές συμπεριφορές πρέπει να είναι ίδιες σε όλες τις χώρες. Προετοιμάζουμε επίσης και μελέτη αντικτύπου που είναι πάρα πολύ δουλειά γιατί πρέπει όλοι, για όλες τις χώρες να έχουμε εμπειρογνώμονες οι οποίοι ξέρουν τι γίνεται, τι δεν γίνεται, τι δεν πρέπει να γίνεται κτλ. Το τελευταίο που θέλω να προσθέσω εδώ είναι ότι πρέπει να ε, βρεθεί και η απαραίτητη χρηματοδότηση για τον εξυγχρονισμό του εξοπλισμού των τελωνίων. Δύο σχόλια θα κάνω για την ιδέα που ακούστηκε στο Κοινοβούλιο ε, να χρησιμοποιηθεί το πρόγραμμα Τελωνία 2020 ε, για την προμήθεια ε, νέου εξοπλισμού σε τελωνία τα οποία έχουν ελλείψεις θετικά βλέπουμε αυτή τη στήριξη που θέλετε να μας δώσετε, αλλά νομίζω ότι το πρόγραμμα Τελωνία 2020 δεν είναι το κατάλληλο πρόγραμμα. Νομίζω ότι είναι καλύτερα τα οι περιφερειακοί πόροι να χρησιμοποιηθούν ε, για, τα, για το σκοπό αυτό. Ε, και οι συνάδελφοι που ασχολούνται με το Περιφερειακό Ταμείο ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι αυτοί οι οποίοι έχουν αρχίσει ήδη να συζητούν το ζήτημα αυτό και έχουν έρθει σε επαφή με τους συναδέλφους των τελωνίων. Τώρα, εάν και μέσα ε, και το πρόγραμμα αυτό, το Τελωνία 2020, συμφωνηθεί ακόμα πιο γρήγορα, τόσο το καλύτερο. Αυτά λοιπόν, δεν θα πω τίποτα άλλο και είμαι στη διάθεσή σας για πιθανές ερωτήσεις. Ωραία. να μη ε, διαθέσουμε ένα δεκάλεπτο για τις ερωτήσεις. Ο κύριος Μπαλντεσάρη είναι υπεύθυνο για το πρόγραμμα για τα τελωνία, είναι εδώ. Ο κύριος Σβάμπ, η κυρία Γκέπχαρτ, η κυρία Βάιλερ ζητούν το λόγο. Η κυρία... ο κύριος Σβάμπ, η κυρία Βάιλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τζούρεκα. Βέβαια καλό θα ήταν να βλέπαμε και τον Επίτροπο, πάντως του ευχόμεθα Περαστικά ευχαριστούμε και για την ωραία ταινία. Δείχνει το μέλλον. Πιστεύω στο μέλλον αυτό και πρέπει όμως να τονίσουμε ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα μέχρι εκεί γιατί στην ε, ανακοίνωσή σας ε, για το Ατελωνία 2020 λέτε ότι χρειάζεται μια στεναρή, ενιαία τελωνιακή ένωση. Συμφωνούμε απόλυτα και ρωτούμε τι κάνει η Κομισιόν για να πείσει τα κράτη-μέλη ότι αυτά που γράφεται εδώ και είναι σωστά θα πρέπει να ακολουθηθούν από τα κράτη-μέλη. Η συγκήτριά μας Κωνσταντς Λεγκρίτ δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα. Ε, εξ ονόματός της λέω ότι ζητάμε να, βρούμε μια, να ρίξουμε μια γέφυρα με την τωρινή κατάσταση και το UCC, τον ενιαίο τελωνιακό κώδικα. Εδώ χρειάζεται ε, μια αισιοδοξία, αλλά ίσως είναι υπερβολικό τον Απρίλιο να καταλήξουμε σε συμφωνία. Θα θέλαμε λοιπόν να βρεθούν, να αναζητηθούν δυνατότητες, αφού το Κοινοβούλιο θα έχει εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες, να ε, συναντηθούμε το Μάιο, ούτως ώστε τον Ιούνιο να έχουμε τον τελωνιακό κώδικα. Και τελειώνω, ε, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο διαφοροποιούνται σε ένα σημείο ε, το δίκαιο περί καταγωγής ε, καλό θα ήταν λοιπόν να στηρίξετε εσείς τη θέση του Κοινοβουλίου γιατί με όλες τις δυσκολίες που έχουμε με τις προτάσεις ε, ε, για τις, ε, τις εκτελεστικές πράξεις εκεί θα έπρεπε να περιοριστούμε στις προτάσεις του Κοινοβουλίου και να μην προχωρήσουμε πέραν αυτών. κυρία Βάιλερ και μετά κυρία Μπαλτασάρη. δεν θα μιλήσω εξ ονόματος της Κιόδους, θα πω κάτι άλλο. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την ε, ωραία παρομοίωση. Ε, Ινδικά χειρίδια, πειραματόζωα και πρωτοπόροι. Δεν το έχω ξανακούσει. Ε, επειδή όμως ε, κάνουμε ανταλλαγή απόψε, δεν θα μιλήσω για τον κώδικα, θα αναφερθώ σε κάτι που μάθαμε χθες σε μια παράλληλη επιτροπή. Η δική Επιτροπή ε, συνεδρίασε και κάποιοι συνάδελφοι, όχι από την Επιτροπή, κάποιοι εμπειρογνώμονες από την επιτήρηση της αγοράς και τα τελωνία, ε, με πολύ γλαφυρό τρόπο ε, μας εξήγησαν ότι η επιτήρηση της αγοράς για εισαγόμενα εμπορεύματα, ε, ειδικά τα μη επιτρεπόμενα ε, wildlife products, ε, ας πούμε ε, ε δέρματα λιονταριών ή ελεφαντοστούν ε, δεν ε, παρακολουθούνται σωστά και υπάρχουν πολλές καταγγελίες και καταδίκες σε άλλες χώρες. Ενώ και βλέπουμε πόσο καλυμμένες είναι οι εισαγωγές του, ελεφαντοστού, του, του ελεφαντόδοντου ε, στην Ευρώπη και μας είπαν ότι ο πέμπτος σε μέγεθος τομέας παραγωγής θα, στο, σε λαθρέα προϊόντα είναι τα προϊόντα άγριων ζώων. Και ρωτώ, επειδή είστε υπεύθυνος και για την επιτήρηση της αγοράς, μπορείτε να το επιβεβαιώσετε αυτό, ότι δηλαδή είμαστε πολύ χαλαροί στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές απαγορευμένων προϊόντων. Γιατί δεν είναι μόνο τεράστια η καταστροφή που υφίστανται οι αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά δεν ε, υπάρχει και προστιθέμενη αξία με αυτόν τον τρόπο που να μπαίνει στην Ευρώπη. Απλώς πρόκειται για ένα έγκλημα, για μια εγκληματική δραστηριότητα. Το λέω γιατί έτυχε να ακούσω από τους ειδικού πώς αντιμετωπίζονται αυτές τις εισαγωγές στην Ευρώπη. Ο κύριος Μπαλτασάρη. Ναι, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να εκφράσω την ευχαρίστησή μου ε, για το βίντεο ε, ε, το οποίο είδαμε και το οποίο μου θύμισε λίγο έτσι των θαλασσών. Πολύ μου άρεσε. Έχει ξεκινήσει λοιπόν λέει η η Κομισιόν ε, μία, ένα νέο πρόγραμμα για, τις, για τα τελωνία 14-20. Οι κύριες ε, προτεραιότητες οι οποίες ανακοινώθηκαν σε αυτό το ε, πρόγραμμα είναι η καταπολέμηση της απάτης, είναι οι τεχνολογικές ικανότητες οι οποίες πρέπει να ενδυναμωθούν, αλλά βεβαίως και η αναθεώρηση του προϋπολογισμού έτσι ώστε να καλυφθούν με καλύτερο τρόπο τα διοικητικά κόστη και στο Συμβούλιο νομίζω ότι προχωράνε με καλό ρυθμό οι εργασίες ε, και είχα τη δυνατότητα να λύσω το πρώτο κείμενο επί του οποίου εργάζονται οι εθνικές αντιπροσωπείες. Επομένως αυτή η νομοθετική διαδρομή έχει ξεκινήσει. Καλά είμαστε σε καλή θέση έτσι ώστε ε, ελπίζω και ευελπιστώ να έχουμε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Τώρα, μια και είστε εδώ, να σας πω, εάν ε, και βάσει της ε, θέσης του Κοινοβουλίου αλλά και βάσει των ε, πολλών γνώσεών σας υπάρχουν ε, κάποια σημεία τα οποία θέλετε να ε, μας πείτε, τα οποία να είναι κρίσιμα, τα οποία να χρειάζονται ιδιαίτερης αντιμετώπισης, τα οποία να αποτελούν έτσι ιδιαίτερο προβληματισμό και σημεία ανησυχίας και για την Κομισιόν και για τους εμπλεκόμενους. Ευχαριστώ. Κυρία Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ξέρετε πρόσφατα συζητήσαμε τον προϋπολογισμό της Ένωσης και είπαμε ότι χρειάζεται ιδίους πόρους η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βασικό θέμα συζητήσεως ήταν ο φόρος χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Για πέστε μας. Σε ποια φάση βρίσκεται η προβληματική. Ακόμη έχουμε μόνο 11 χώρες οι οποίοι θέλουν να προωθηθεί το, το, το, η υπόθεση αυτή. Τι γίνεται, πώς έχει η κατάσταση. Ναι, ναι, απαντήστε αυτές τις ερωτήσεις, αν θέλετε. Και ίσως μπορέσουμε, αν έχουμε χρόνο, να κάνουμε και άλλο ένα γύρο ερωταπαντήσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω ότι δεν είναι αδικαιολόγητη η αισιοδοξία μου. Εγώ εξεπλάγην θετικά από την ταχύτητα με την οποία έγιναν οι χειρισμοί πολύ σύνθετων αλλά και πολιτικά επίμαχων θεμάτων σε τεχνικό επίπεδο. Ε, αυτών που έχουν σημασία για τα τελωνία. Κινήθηκαν με ταχύτητα και τα δύο θεσμικά όργανα. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Γιατί υπάρχει συμφωνία ότι και οι δύο θέλουν να κάνουν το καλύτερο για την Τελωνιακή Ένωση. Ελπίζω να τηρήσουμε την προθεσμία του Απριλίου και πολύ γρήγορα να φτάσουμε ε, στην ε, συμφωνία. Θέλουμε αυτή τη γεφύρωση να την διαμορφώσουμε έτσι, ούτως ώστε να είναι αρκετή για το σωστό χειρισμό του θέματος. Δεύτερον, ε, εξαγωγές. Σε αυτό το τομέα δεν προτιθέμεθα να αναλάβουμε πρωτοβουλία. Δηλαδή, δεν θέλουμε το τέρας του Λοχνές ε, να το προκαλέσουμε. Ε, άλλωστε δεν, ε, ε, δεν μας μόλυνε εμάς με τα αυγά του, δεν αναπαρήχθη. Τώρα για την επιτήρηση της αγοράς, μαζί με τους συναδέλφους από την εσωτερική αγορά και τις επιχειρήσεις και το εμπόριο προσπαθούμε να ε, στήσουμε ένα σύστημα πιο αποτελεσματικό. Εδώ χρειαζόμαστε μεγάλη υποστήριξη από το Κοινοβούλιο. Εν τω μεταξύ υπάρχει η τάση να μην εξοπλίσουμε επαρκώς τους μηχανισμούς επιτήρησης της αγοράς. Ε, θα υπήρχε, υπάρχει ε, τραπεζική εποπτεία αποτελεσματική. Όλες οι άλλες εποπτείες ε, υποστελεχώνονται και δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης ότι οι τελωνιακές αρχές έχουν να αντιμετωπίσουν ε, συνεχώς αυξανόμενες ροές εισαγωγών, πράγμα που δυσχεραίνει όλο και περισσότερο τους ελέγχους. Γι' αυτό προσπαθούμε να εισαγάγουμε ένα σύστημα που θα στηρίζεται στην αξιολόγηση του κινδύνου. Τώρα για το δεύτερο ερώτημα, τις ε, εισαγωγές ε, απαγορευμένων προϊόντων ζωικών. Ξέρουμε ότι η Συμφωνία Προστασίας της Ουάσιγκτον σε μεγάλο βαθμό έχει ενσωματωθεί στο διεθνές δίκαιο και έτσι ε, θα πρέπει τα δικαστήρια να λαμβάνουν υπόψη τις διατάξεις αυτές. Η τελωνιακή έχουν καθήκον να κατάσχουν τα απαγορευμένα εισαγόμενα προϊόντα και οι δράστες που έκαναν την απόπειρα να εισάγουν τα προϊόντα να διωχθούν. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι χρειάζεται εναρμόνιση των κυρώσεων, ούτως ώστε να μην μπορεί κανείς να διαλέγει το πιο ευνοϊκό δικαστήριο για να γλιτώνει μετά από τις εισαγωγές ε, ελεφαντόστου και άλλων τέτοιων παράνομων προϊόντων στην Ευρώπη. Όλα αυτά εμείς τα ε, προσεγγίζουμε με μεγάλη σοβαρότητα, αλλά είμαστε αντιμέτωποι με μια δραστηριότητα η οποία ε, είναι εν μέρη τόσο άτυπα οργανωμένη που δύσκολα εντοπίζεται και διώκεται. Πάντως αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω πόσο ε, μεγαλύτερες είναι αυτές οι εισαγωγές στην Ευρώπη σε σχέση με άλλες περιοχές του κόσμου. Πάντως θα κοιτάξω να βρω τις πληροφορίες που θέλετε και να σας τις στείλω. Κύριε Μπαλτεσάρε, είμαι πολύ ευτυχής που ακούω ότι προχωρήσατε τόσο πολύ και είσαστε έτοιμοι για την έναρξη του τριμερούς διαλόγου. Πολύ χαίρομαι που το ακούω. Ομολογώ ότι δεν είμαι σε θέση να ε, καταδείξω κάποια συγκεκριμένη διαφορά ή κάποιο επίμαχο θέμα στις προτεραιότητες οι οποίες είναι ξεκάθαρες τουλάχιστον για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι δύο ειδών. Πρώτον, να επιτρέψουμε να ε, λειτουργούν οι τελωνιακές υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη και να έχουμε τεχνολογία της πληροφορίας που χρειάζονται για τον ε, ενωσιακό τελωνιακό κώδικα. Αυτό είναι πολύ σημαντικά. Είναι πολύ φιλόδοξο το σχέδιο της ανάπτυξης της ε, τεχνολογίας της πληροφορίας. Νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητα που έχουμε σήμερα. Η κυρία Τούνφον Χόνσταν για τους ίδιους πόρους και το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Τώρα εξετάζεται το θέμα αυτό μεταξύ των κρατών μελών που τάχθηκαν υπέρ τη ενισχυμένη συνεργασία και τα οποία είναι 11 επί του παρόντος. 11 κράτη-μέλη το κάνουν αυτό. Δεν προσθέθηκε κανένα ακόμα. Δεν μπήκε στο ring άλλο. Αλλά δεν αποκλείεται να συμβεί και αυτό. Πάντως τώρα είμαστε στα σπάργανα της διαδικασίας αυτής γιατί πρόσφατα υπέβαλε τη νέα πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τώρα την μελετούν ε, με κάποια αρχική αμηχανία τα κράτη-μέλη. Και συνεχίζω. Αυτό που θα ήθελα να κάνουμε τώρα είναι να δούμε την πιο μακροπρόθεσμη προοπτική που θα μας κρατήσει απασχολημένους και μας και σας στα τελωνία το επόμενο διάστημα. Εμείς θέλουμε μία ασφάλεια ε, που θα λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο και θα ε, βελτιώνει την ε, ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Θέλουμε να επικεντρωθούμε στην διαχείριση του κινδύνου και θα εντοπίσουμε κενά και λήψεις στα κράτη-μέλη και θα τα αντιμετωπίσουμε και θα είμαστε πολύ ευτυχείς αν από μας υποστήριζε η η Επιτροπή σας εδώ. Τώρα, στο τομέα της ασφάλειας και στο θεματολόγιο της ασφάλειας υπάρχουν πολλά επιμέρους θέματα, όπως αεροπορική, ναύλη, φορτία. Και έγινε ένα πιλωτικό πρόγραμμα μαζί με τις Ηνωμένε Πολιτείες και άλλους αεροπορικούς αερομεταφορείς και μάλιστα ε, μεταφορής express. Ολοκληρώθηκε αυτό το πιλωτικό στο τέλος του έτους και τώρα ε, στηρίζουμε τις ε, διαβουλεύσεις μας επί των αποτελεσμάτων του πιλωτικού προγράμματος για να ξεκαθαρίσει το σύστημα και να δούμε τι δεδομένα χρειαζόμαστε πριν φορτωθούν τα εμπορεύματα στο αεροπλάνο το καλό είναι ότι έχουμε πολύ καλή συνεργασία και από τους, ε, τις Γιατί βεβαίως και εκείνοι ε, ενδιαφέρονται να μην κρύγνονται τα αεροπλάνα τους πάνω από τον ωκεανό, αν φορτωθούν εκρηκτικά. Τώρα, πώς θα αντιμετωπίσουμε τις χώρες από τις οποίες προέρχονται τα φορτία αυτά. Θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία και πρέπει να βρούμε σοβαρούς και αξιόπιστους εταίρους. Έτσι θα μπορέσουμε να υπογράψουμε με τις ΗΠΑ μια συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης που θα αναγνωρίζει τους εξουσιοδοτημένους οικονομικούς μας επιχειρηματίες ε, που θα δραστηριοποιούνται στις Ηνωμένε Πολιτείες. Έτσι θα έχουμε και ανταλλαγή δεδομένων και ένα εργαλείο ε, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων που θα αφορούν τα φορτία, τους ναύλους. Ε, και προς Ανατολάς ε, όμως έχουμε ενδιαφέροντες γείτονες, Ουκρανία, Μολδαβία, Ρωσία. Με αυτές τις χώρες θέλουμε να προχωρήσουμε το θεματολόγιο της ασφάλειας, το οποίο είναι σημαντικό για να έχουμε εμπορικούς δρόμους ασφαλή, να γίνεται διαχείριση του κινδύνου, να καταπολεμούνται οι απάτε και να υπάρχει και εξυγχρονισμό των τελωνίων. Και εκεί. Πολλές χώρες υποφέρουν γιατί υπάρχουν μεγάλες ουρέ λεωφορείων, ε, όχι λεωφορείων, φορτηγών που πρέπει να εκτελονίσουν τα εμπορεύματά τους ε, και ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο πρόβλημα τώρα που πάμε να βρούμε συμφωνία με τους Ρώσους και είναι δύσκολο. Τώρα λένε δεν είμαστε πια μόνο η Ρωσία, είμαστε μαζί με το Καζαχστάν και τη Λευκορωσία σε τελωνιακή ένωση. Περιπλέκεται το θέμα και υπάρχει κάποια προθυμία να ε, αρχίσουν επίσημες σχέσεις με αυτήν την τελωνιακή ένωση. Αυτό δυσκολεύει τα πράγματα. Μας παίζουν λίγο τώρα παίζουν λίγο πινκ-πονγκ μαζί μας. Καμιά φορά φορούν το καπέλο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, άλλες φορές της ε, Τελωνιακής Ένωσης με τις χώρες αυτές και αυτό δυσκολεύει τα πράγματα. Όμως αυτό αντισταθμίζεται διότι υπάρχει η ιδέα αυτή των εξανατολών γειτόνων να βελτιώσουν τις μεταφορές και τον εκτελονισμό. Η Κίνα είναι πολύ σημαντική επίσης ε, ε, στο εμπόριο και επιτελούμε πρόοδο στην τελωνιακή συνεργασία, την ε, επιβολή δικαιωμάτων διανοητικής ε, ιδιοκτησίας και άλλα. Προσπαθούμε να αναπτύξουμε προγράμματα και έχουμε, προοδεύουμε. Τώρα, για το συνολικό θέμα της διακυβέρνησης της Τελωνιακής ε, Ένωσης, έχουμε εδώ ένα θέμα ακόμα. Έχουμε μια Τελωνιακή Ένωση, η οποία είναι σχεδιασμένη με βάση την πραγματικότητα της δεκαετίας του 50 και δημιουργήθηκε στα πλαίσια του περιβάλλοντος που επικρατούσε τη δεκαετία του 60. Ενώ τώρα έχουμε αυξήσει όχι μόνο τον αριθμό των μελών της Τελωνιακής Ένωσης, αλλά άλλαξε και το επιχειρηματικό περιβάλλον άρδιν. Και ακόμα εμείς είμαστε αντιμέτωποι με την ίδια κατάσταση και έχουμε 27, σύντομα 28 μεμονωμένα κράτη-μέλη, τα οποία οργανώνουν τις δικές τους θελωνιακές τους ε, αρχές, πράγμα που μειώνει την γενικότερη αποδοτικότητα του συστήματος. Εμείς τώρα κάνουμε μια αξιολόγηση, έχουμε το πρώτο, το, την πρώτη ε, ανακοίνωση, την οποία... Ε, υποβάλαμε και περιμένουμε τι αντιδράσει του Συμβουλίου αλλά και από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και θα ήμουν ευτυχής αν και το Κοινοβούλιο θα μπορούσε παρακαλώ να ε, εξετάσει λίγο το έργο αυτό γιατί είναι ένα θέμα όπου έρχονται και μας βρίσκουν οι εμπλεκόμενοι και μας λένε μιλήστε και με τους βουλευτές που ξέρουν ε, τα θέματα αυτά. Αυτά λοιπόν τα τελωνιακά, οι πρωτοβουλίες και για τον ΦΠΑ τώρα δύο λόγια πολύ γρήγορα. Τώρα δουλεύουμε. Πάμε να εξυγχρονίσουμε το σύστημα του ΦΠΑ γενικότερα, αλλά έχουμε και κάποια επιμέρους θέματα που είναι πιο κατεπήγοντα. Ε, ένα πράγμα που θέλω να σας πω είναι το θέμα των συντελεστών ΦΠΑ και οι μονοπευθυντικές θηρίδες που είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τις μικρές επιχειρήσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους συντελεστές, το ποσοστό του ΦΠΑ, το θέμα είναι ότι είναι κατεπήγον το θέμα εν ώψη της εξέλιξης της ψηφιακής εσωτερικής αγοράς. Γιατί όταν ο κατάλογος των προϊόντων που θα είναι επιλέξιμα για μειωμένο φορολογικό συντελεστή θα είναι έτοιμος, όταν ο κατάλογος θα είναι έτοιμος, κανείς, βέβαια με ελάχιστε εξαιρέσεις, κανείς δεν θα είναι έτοιμος για ένα ηλεκτρονικό σύστημα. Τώρα έχουμε ένα κατάλογο ε, αντικειμένων που είναι επιλέξιμα για ηλεκτρονικό εμπόριο, ε, που ε, είναι προϊόντα πολιτιστικού περιεχομένου. Τώρα τι είναι αυτό είναι λίγο γενικό λόγο. Αλλά τα ηλεκτρονικά βιβλία θεωρούνται υπηρεσία με βάση την προσέγγιση αυτή και υπόκειται στον ε, πλήρη φορολογικό συντελεστή. Θεωρούμε ότι δεν είναι καλή λύση αυτή. γιατί προϊόντα που εξυπηρετούν με παρόμοιο τρόπο τον καταναλωτή πρέπει να αντιμετωπίζονται με παρόμοιο τρόπο και από εμά. Αλλά εμείς θέλουμε να υποβάλουμε μια πρόταση που θα συμπεριλαμβάνει και την αρχή αυτή που σας είπα ότι ό,τι εξυπηρετεί με παρόμοιο τρόπο τον καταναλωτή πρέπει να αντιμετωπίζεται με, τον ίδιο τρόπο και πρέπει να λάβουμε υπόψη μα και την εξέλιξη τη τεχνολογία. Γιατί μπορεί να προκύψουν και άλλα πράγματα καινούρια που δεν τα ξέρουμε σήμερα και τα οποία μπορεί να επηρεάσουν πολύ την αγορά στο μέλλον. Αυτή είναι μια πρόταση λοιπόν που ακόμα ετοιμάζουμε για να την έχουμε έτοιμη τέλος του χρόνου. Θα την έχετε δηλαδή ε, την πρόταση μπροστά σας πριν από τις εκλογές και καλή επιτυχία σας εύχομαι. Το άλλο είναι η μόνο απευθυντική θηρίδα, ε, την ηλεκτρονική πια γιατί όταν ο ΦΠΑ θα εισπράτεται αυτό είναι για τις μικρές επιχειρήσεις να μην έχουν περίπλοκο σύστημα για την υποβολή του ΦΠΑ αυτό θα γίνεται σε μόνο απευθυντική θηρίδα ε, εδώ ακολουθούμε τα χρονοδιαγράμματα 1η Φεβρουαρίου του 2015 θα πρέπει να είναι λειτουργικό το σύστημα το καινούριο και προς το παρόν βλέπουμε και τα κράτη-μέλη να θέλουν να αφιερώσουν επαρκείς πόρους για την δημιουργία και την εξάπλωση του συστήματος. Τεράστιο καθήκον βέβαια να το εξηγήσουμε στα 23 εκατομμύρια μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη και να τους εξηγήσουμε ότι θα ωφεληθούν από το καινούριο σύστημα. Αυτά είναι οι, τα δύο, οι δύο άμεσες προτεραιότητες που ήθελα να σας υποβάλω και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι είναι ε, πολλοί που ενδιαφέρονται ε, για, την, ε, για το χαμηλότερο ΦΠΑ σε ηλεκτρονικά βιβλία. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να μιλήσει για το χαμηλότερο ΦΠΑ ή για τα Kindle και τα ηλεκτρονικά βιβλία ή τη μόνο απευθυντική θηρίδα. Να πω μόνο ότι όχι μόνο η Γερμανία, αλλά βεβαίως και πολλά άλλα κράτη-μέλη δεν έχουν συνεκτικό σύστημα για τον ε, μειωμένο ή όχι μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ. Κομμένα λουλούδια, μειωμένος. άλλα, οι τρόφιμα, ζωοτροφές, νομίζω και αυτά είναι μειωμένα. Οι πάνες για τα μωρά όχι. Πάντω υπάρχουν διαφορέ, δεν υπάρχει συνεκτικό σύστημα, ομοιόμορφο. Να ειδού λοιπόν λαμπρή ευκαιρία, αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πανεξετάζει το σύστημά της, χρυσή ευκαιρία να το κάνουν αυτό και τα κράτη-μέλη. Γιατί ξέρω ότι ε, σε εμά υπάρχει αυτή η συζήτηση. Αλλά πρέπει να προσέξουμε να μην ε, γίνει ε, ως, λένε συνήθως ότι από τις Βρυξέλλες έρχονται οι υψηλοί συντελεστές και οι μειωμένοι συντελεστέ για του καταναλωτέ προέρχονται από τα κράτη-μέλη. Όχι, θα πρέπει να είναι μια συνεκτική συζήτηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεύτερον, δεν μα είπατε τίποτα για, τον, για το, ότι απάτες με τον ΦΠΑ που στην Ευρώπη δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να το προσέξουν αυτό το θέμα περισσότερο γιατί έτσι θα αυξήσουν και τα έσοδα για τον προϋπολογισμό. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να περιορίσει, να ανασχέσει αυτές τις τεράστιες απάτες με τον ΦΠΑ. Θέλει κάποιος άλλος να σχολιάσει. Παρακαλώ. Κυρία Βάιλερ, αν η Γερμανία δεν έχει συνεκτικό σύστημα στην εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή, αυτό οφείλεται σε δύο λόγους. Πρώτον, ο κατάλογος των εμπορευμάτων ή υπηρεσιών που είναι επιλέξιμα για το μειωμένο συντελεστή πρέπει να ε, αποφασιστεί ομόφωνα από όλα τα κράτη-μέλη. Και εδώ υπάρχουν ορισμένα, ε, ε, ορισμένες αναντιστοιχίες. Ε, το άλλο, άλλος λόγος που είναι πολύ πιο μεγάλος και σοβαρός, κανείς δεν αναγκάζει τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν μειωμένο συντελεστή καταρχήν και ο κατάλογος των προϊόντων που ε, υπόκεινται σε μειωμένο ε, συντελεστή είναι θέμα τη εθνικού δικαίου. Οπότε αυτές τις παρατηρήσεις θα πρέπει να τις απευθύνεται μάλλον προς το Γερμανό νομοθέτη, ο οποίος θα μπορούσε να φροντίσει για μεγαλύτερη συνέπεια. Και εμείς το επιχειρούμε μέσα από την πρότασή μας για τους διαφορετικούς φορολογικούς συντελεστές, ούτως ώστε να βρούμε ένα πιο διεθνές σύστημα αν θέλετε. Αλλά όταν υπάρχουν εθνικές διαφορές υπάρχουν και ε, διαφορετικά αποτελέσματα. Είχαμε και ε, μια συζήτηση με Γάλλους επιχειρηματίες που μας είπαν ότι πολλές φορές ε, σε σχέση με το σκάνδαλο με το κρέας αλόγου και τους συντελεστές και μας είπαν ότι θα πρέπει να το προσέξουμε αυτό γιατί μπορεί να επηρεάσει την κατάσταση. Η επιλογή πάντως των προϊόντων που υπόκεινται σε μειωμένο φορολογικό συντελεστή, η απόφαση αυτή είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Και μόνο ο τομέας επιλογής αυτών των ε, προϊόντων είναι αντικείμενο που ρυθμίζεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς πάντως προσπαθούμε τώρα να εναρμονίσουμε το σύστημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που ακούσαμε. Μπορέσαμε και εμείς ε, να θέσουμε ερωτήσεις και εσύ μας έδωσε συγκεκριμένα σχέδια της ε, Κομισιόν περιμέναμε ε, από καιρό έτσι, τα πράγματα αυτά, τις αποσαφηνήσεις ε, και πολύ ωραίο και το φιλμάκι. Μήπως μπορούμε να το φορτώσουμε και μόνοι μας από το YouTube, θα δούμε. Για τον ΦΠΑ ε, τα στοιχεία αυτά τα οποία αναφέραμε και αυτή η θηρίδα η ενιαία είναι πολύ σημαντικά θέματα για τα οποία και εμείς δουλεύουμε πολύ. Ευχαριστούμε που ήρθες, που μας μίλησες για τα ζητήματα αυτά. Πολύ βοήθησε τη συζήτηση. Και βεβαίως ε, τις καλύτερες ευχές μας στον Επίτροπο Σεμέτα ε, και βεβαίως να του ευχηθούμε ταχεία ανανάρρωση. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Να πω ότι το βίντεο αυτό είναι διαθέσιμο σε 23 γλώσσες. Uh, Πρόεδρος, λοιπόν, συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διατάξεως του απογεύματος. Είναι η μελέτη των συμβαστικών τροπολογιών επί της εκθέσεως Γκαρθές Ραμών. Νέα ατζέντα για την ευρωπαϊκή πολιτική καταναλωτών. Βλέπω την κυρία Κανιέτε που είναι εδώ, ο κύριος Μέντες, ο οποίος ενδεχομένω εκπροσωπεί... Ε, το... Α, όχι, όχι, δεν εκπροσωπείται κανέναν. Η κυρία Ρούλη είναι εδώ. να ζητήσω συγγνώμη στην Επιτροπή, γιατί στις 4.30 πρέπει να συναντήσω τον κύριο Βαν Ρόμποη, τον πρόεδρο του Συμβουλίου, να συζητήσουμε για την ε, ε, για την ένταξη των θεμάτων ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς ε, στις πολιτικές και στρατηγικές του Συμβουλίου. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να φύγω. Ε, πρέπει να σας πω ότι τον ενδιαφέρουν πάρα πολύ όλα αυτά που κάνουμε εδώ, κυρίως αυτά που κάνουμε για την ψηφιακή οικονομία. Βεβαίως θα σας κάνω μετά αναφορά. Η κυρία Βάιλερ συμφώνησε να προεδρεύσει από τις 4 και 25 περίπου. Μήπως προτιμάτε όμως να ξεκινήσετε από τώρα έτσι ώστε να γίνει πιο εύκολα. Α, και επίση, αν έρθετε από τώρα να προεδρεύσετε, εγώ θα βάλω και το καπέλο του σκιώδου συγητού για το θέμα αυτό τη ημερησία διάταξη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, να μας πει ο κύριος Γκαρθές Ραμών ε, την πρώτη του, τα πρώτα του σχόλια και μετά συνεχίζουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, Los trabajos relativos a la nueva agenda del consumidor. Οι εργασίε προχωρούν όσον αφορά για το κύριο χάρτη δικαιωμάτων του καταναλωτή. Κάτι πάρα πολύ ε, απαραίτητο. Ε, νομίζω το αποτέλεσμα θα μα δικαιώσει, θα είναι άριστα και πότε πρώτα πρώτα να ευχαριστήσω για τι προσπάθειε που κατέβαλαν οι ηγητέ. τα είπαμε επανειλημμένα, οπότε και έτσι μπορέσαμε να εξεύρουμε σημεία συμφωνίας και να βελτιώσουμε τις προτάσεις. Επίσης, θα πρέπει να ευχαριστήσω για την υποστήριξή τους ε, όλους τους συνεργάτες μας. Οπότε και αυτή η νέα ατζέντα θα βελτιώσουμε όλο ένα και περισσότερο. 213 είναι οι πολυθήσεις τροπολογίες όσον αφορά το αρχικό κείμενο. Και τελικά καταλήξαμε εις 21 συμβαστικές τροπολογίες. Εκείνες που καλύπτουν πάνω από 90 εκ των αρχικά υποβληθισών τροπολογιών. Και οπότε έτσι θα είμαστε εις θέση να πετύχουμε την σύνεση εκείνη που θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε ευκολότερα. Αυτές λοιπόν οι συμβαστικές τροπολογίες αναδεικνύουν το πόσο χρειάζεται να βελτιώσουμε την ενημέρωση, κατάρτιση τελικά των καταναλωτών, εκτός από κάποιες οικονομικές πτυχές. Αυτό να γίνεται λοιπόν με διάφορο τρόπο, με πάγιο τρόπο, με συγκρισιμότητα, με αξιοπιστία, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε ασφάλεια, ανιχνευσιμότητα και αυθεντικότητα των προϊόντων. προϊόντων συγγνώμη. να είναι σίγουρη η κατάσταση, ούτως ώστε να μην εξαπατώνται οι καταναλωτές. Και όλα αυτά στο γενικότερο νομικό πλαίσιο με ανεξάρτητη αξιολόγηση. Οπότε και να μπορούν να έχουν σε αυτές τις εκτιμήσεις εμπιστοσύνη καταναλωτές. Επίσης, με αυτές τις μελλοντικές τροπολογίες θέλω να εμείνουμε στο πόσο χρειάζεται να αποφύγουμε κάποιες πρακτικές και κάποιες ρήτρες καταχρηστικές και, και, και ώστε να προστατεύσουμε τους ε, παγιδευθέντες ε, καταναλωτές σε διάφορα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Αυτό έρχεται να σχετιστεί με κάποια φαινόμενα τα οποία γύρω-γύρω λόγω χώρα λόγω της χρηματοοικονομικής κρίσης την οποία περνάμε τα τελευταία χρόνια. Οπότε και όλο ένα και περισσότερος κόσμος πλήσεται από αυτό το φαινόμενο. Γι' αυτό και αξίζει να προσέξουμε ιδιαίτερα το πρόβλημα αυτό σε αυτή την νέα ατζέντα. Και τώρα και στις πιο εξελιγμένες μορφές. Οπότε έχουμε τους πιο ευάλωτους ε, καταναλωτές που θα πρέπει να τους προσέξουμε ιδιαίτερως. Σε μεταφορές, σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, σε ενέργεια, στις νέες τεχνολογίες ενημέρωσης και πληροφόρησης. Οπότε έτσι έχουμε εκεί στις υπερχές τροπολογίες ένα λογαριασμό πληρωμής που μπορεί να λειτουργήσει με αξιόπιστο και ασφαλή τρόπο. Όπως είπαμε λοιπόν, το σοβεί η κρίση, η χρηματοοικονομική και γι' αυτό οι ανισότητες όλο ένα και αυξάνονται. Και μεταξύ χωρών και μέσα στην ίδια τη χώρα, οποιαδήποτε χώρα. Οπότε αυτό το βιώνουν πάρα πολύ αρνητικά οι καταναλωτές. Οπότε και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι και να φροντίσουμε και την κοινωνική πτυχή της ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Αναφίβολα, η επίλυση των διαφορών. Ε, είναι θέμα πολλών τροπολόγιων. Θα πρέπει να είναι αποτελεσματική, θα πρέπει να είναι ταχεία, θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη η δικαιοσύνη ή τόσο τα όργανα τα δικαιοδοτικά και οπότε και γι' αυτό η Επιτροπή προτείνει κάποιο ειδου ε, μηχανισμούς ε, συλλογικών προσφυγών και επίσης τροπολογίες, λέμε το πόσο χρειάζεται, να υπάρχουν κάποιες εγγύσεις για τις διασυνολογικές αλλαγές. Όπου χρησιμοποιούνται ευρέως στο εμπόριο. Τώρα, όσον αφορά τον ρόλο των ενώσεων καταναλωτών, ε, θα πρέπει αυτές τις ενώσεις να τις ε, βοηθήσουμε, να τις υποστηρίξουμε και επίσης στις τροπολογίες τονίζεται ότι θα πρέπει να βρεθούν κάποιοι τρόποι, ώστε αυτές οι ενώσεις καταναλωτών να επιτελούν το έργο τους με καλύτερο τρόπο. Εντάχει λοιπόν και συνθετικά αυτό είναι το περιεχόμενο των θεσμών τροπολογιών. Και περιμένω να μου πούν τη γνώμη τους και και έτσι να μπορέσουμε να βάλουμε στις τελευταίες πινελιές στο στην έκθεσή μας. Η Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κάνη η κυρία Ρίουλε, ο Μάλγκον Χάρμπερ. Οι τρεις σκιώδεις ζητούν το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πολύ αποτελεσματική συνεργασία που είχε με μας τους σκιώδεις εισηγητές. Ε, κατάφερε να επιτύχει μεγάλο βαθμό συνένεσης και έβαλε και τις δικές μας απόψεις στην έκθεσή του πρέπει να πω ότι έλαβε υπόψη του τα περισσότερα πιο σημαντικά ε, σημεία του ΕΛΚ. Ε, είχαν υποβληθεί πάνω από 200 τροπολογίες ε, και επ' αυτών είχαμε συμφωνία επί συμβιβαστικών τροπολογιών. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι έχουμε εκφράσει και επικριτική στάση απέναντι στην έκθεση της Κομισιόν θα κάνουμε και συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να διασφαλιστεί και οι προσαναλωτών ε, και οι οικονομικές δραστηριότητες. Θα τις υποβάλουμε με την ελπίδα ότι θα τις λάβει υπόψη της ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκθεση αυτή δεν αφορά μονάχα τους καταναλωτές και τα δικαιώματά τους, αλλά ε, ε, αναφέρεται και στις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις ε, πρέπει να γνωρίζουν τα δικαιώματα των καταναλωτών και να λαμβάνουν υπόψη τους αυτά τα υψηλά επίπεδα απαιτήσεων όσον αφορά τους καταναλωτές και βεβαίως αντιστοίχως να προσαρμόζουν τις υπηρεσίες τους. Τέλος, να πω ότι είμαι βεβαία ότι σε μερικές εβδομάδες θα εγκριθεί η έκθεση αυτή με πλειοψηφία στην Επιτροπή μας. και θα είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως, όχι μονάχα τον εισηγητή, αλλά και την κυρία Ρούιλε ε, και τους άλλους συναδέλφους και τον Μάλκον ε, που βοήθησαν στην ολοκλήρωση της έκθεσης αυτής. Ε, και τελευταία να ευχαριστήσω την Γραμματεία και του, της και τους βοηθούς μας που δούλεψαν σκληρά έτσι ώστε να επέλθει συμφωνία όσον αφορά την τελική εκδοχή αυτού του εγγράφου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ η κυρία Ρούλα για τους πρασίνους. Προχωράμε πιο γρήγορα από ό,τι φανταζόμουν. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω για την εξαιρετική δουλειά και τον εισηγητή και τη γραμματεία. Η εργασία αυτή και οι συμβιβαστικέ τροπολογίε ήταν τα σημαντικότερα. Ε, στέφθηκαν από επιτυχία και ευχαριστούμε. Γιατί με τι συμβιβαστικέ νομίζω ότι θα έχουμε την πλειοψηφία στην Επιτροπή μα και θέσαμε σημαντικές προτεραιότητες γιατί με τη βαθιά οικονομική κρίση πρέπει και εμείς να ε, ασκούμε μια πολιτική αποτελεσματική. Ο κύριος Χάρμπορ, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συμφωνώ με τους συναδέλφους και νομίζω ότι επιτελέσαμε σημαντική πρόοδο χάρη στην συνεργασία του εισηγητή του Γιατί επικεντρωθήκαμε στην έκθεση αυτή στην υποστήριξη και ανάδειξη της σημασίας του θεματολογίου των καταναλωτών που ήθελε και η Κομισιόν. Νομίζω ότι ευθυγραμμιστήκαμε σε μεγάλο βαθμό και οι συμβιβαστικές τροπολογίες των και οι προπολογίες των συναδέλφων προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκαν. Ευχαριστώ τους Κιώδης γιατί, που ήταν συνεργάσιμοι, γιατί είναι καλές οι συμβιβαστικές τροπολογίες. Δεν λέω σε αυτό το στάδιο ότι η ομάδα μου θα τις υποστηρίξει όλες, αλλά νομίζω ότι τις περισσότερες θα τις υποστηρίξουμε. Επειδή είμαστε μικρή ομάδα, ε, μπορώ να πω ότι θα στηρίξουμε την ε, έκθεση συνολικά. Κάποιες ε, τμηματικές ψηφοφορίες θα ζητήσω. Τώρα, ορισμένα σημεία που είχαμε κάποιες διαφωνίες. Ε, μία αιτιολογική σκέψη που κάλυψε τροπολογίες από την Επιτροπή Μεταφορών προκάλεσε το ενδιαφέρον. Η Επιτροπή Μεταφορών ήδη έχει περάσει από αυτή τη διαδικασία και τώρα εφαρμόζει πολλά δικαιώματα για τις μεταφορές επιβατών. Ε, υπάρχουν λοιπόν κάποιες ε, αιτιολογικές σκέψεις που φαίνονται λίγο επαρχαιωμένες. Πάντως, ε, αν επιμένει η Επιτροπή Μεταφορών δεν θα πούμε όχι, παρόλο που μας φαίνεται περίεργο. Ε, επίσης, Στην συμβιβαστική 18 ε, αναφέρεται κάτι παράξενο. Η συνεργασιακή κατανάλωση, η συνεργατική. Να μελετήσουμε νέες μορφές κατανάλωσης καλούμεθα εκεί. Αλλά δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Τι είναι. Πάντως, ε, καλό είναι να το ε, εξερευνήσει αυτό η Κομισιόν. Τι είναι αυτό το collaborative consumption. Επίσης, ε, στη συμβιβαστική 10. Η 10 μου φαίνεται ότι είναι ε, πολύ επεμβατική και δεν περιορίζεται σε κάποιες ε, γενικές διατάξεις όπως θα θέλαμε σε σχέση με τη συλλογική προσφύγη. Πάντως γενικά μου φαίνεται ότι φτιάξαμε καλή έκθεση εδώ και όταν θα φτάσουμε στην τελική ψηφοφορία θα ψηφίσουμε υπέρ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Άλλοι σκιώδε δεν παρευρίσκονται αυτή τη στιγμή. Πριν δώσω το λόγο στην Κομισιόν, θέλει κάποιος άλλος βουλευτής να λάβει το λόγο. Συμφωνούν όλοι. Δηλαδή φτάσαμε να μπορούμε να ψηφίσουμε ήδη από αύριο. Μην ανησυχείτε, μην ανησυχείτε, τον άλλο μήνα θα ψηφίσουμε. Η Κομισιόν έχει το λόγο τώρα. Δύο εκπρόσωποι της Κομισιόν είναι παρόντες. θα... Α, διαβουλεύεστε ακόμα η Κομισιόν. Είναι οι κύριοι Μίκολ και Μανφρέντι, κύριος και κυρία. Ζήτησαν το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ θετική στην τροπολογία και ε, ιδίως άπαξ και ξεκαθαρίζεται η σχέση με την νέα ατζέντα για τον καταναλωτή. Ακριβώ έτσι όπω έχει τοποθετηθεί, θεωρούμε ότι αυτή η αποσαφήνιση είναι πάρα, πάρα πολύ χρήσιμη. Αυτό που θέλω να σα πω, ε, το πω ταχαίω, διότι πρώτα-πρώτα θέλω να σα πω κάτι για την ασφάλεια των προϊόντων. Μια που στι τρει τροπολογίε έχουμε κάτι το οποίο συνδέει την αυθεντικότητα με την επικίνδυνοτητα του εμπορεύματος του αγαθού. Και για μας όμως ε, πρόκειται εδώ περί δύο διαφορετικών ενιών. Από τη μία μεριά έχουμε τα επικίνδυνα ε, αγαθά, την, από την άλλη μεριά έχουμε τις απομίσεις, Μπορεί να υπάρχει κάποια επικάλυψη, αλλά πρόκειται για ε, μια διατύπωση εδώ που είναι ευρετάτη τόσο πολύ τελικά δεν, είναι το θέμα τόσο μεγάλο, τόσο τρομερό. Το θέμα είναι η επισήμανση, η ταυτοποίηση του προϊόντος, ε, εκεί που λέμε και για την ενχρησιμότητα. Τώρα, όσο αυτές τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, μας ε, ανέφερε ο εισηγητής ε, το θέμα των συμβουλών των αντικειμενικών, ανεξαρτήτων. Κάνα πρόβλημα και έχουμε άλλωστε και την πρόταση MIFID της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου και σας παραπέμπω. Τώρα έχουμε ε, κάποιες παρατηρήσεις όσον αφορά τις πληροφορίες οι οποίες θα πρέπει να παρέχονται και με λειτουργική μορφή και με άλλες μορφές. Είπαμε εδώ υπάρχει διάζευξη. Είτε έτσι είτε αλλιώ να αναφέρεται. Είτε είτε. Ιδίω όσον αφορά τι πληροφορίε, οι οποίε θα πρέπει να παρέχονται και να είναι προσβάσιμε συνεχώ. Τώρα, όσον αφορά την πρωτοβουλία για τον ε, λογαριασμό, τον τραπεζικό λογαριασμό. Μας αρέσει επίσης αυτό το οποίο προτείνεται αυτή η πρωτοβουλία, όμως ίσως θέλει η Επιτροπή σας να παραπέμψει στους τρεις πυλώνες αυτής της πρωτοβουλίας. έχουμε την πρόσβαση στον ε, τραπεζικό λογαριασμό, αλλά και το θέμα της ε, διαφάνειας, όπως επίσης και το switching ε, αυτή η μετάβαση, α πούμε, το switching, που είναι όλα πάρα πολύ σημαντικά για τον καταναλωτή. Και τα τρία πολύ σημαντικά. Τώρα, όσον αφορά αυτές τις συλλογικές προσφυγές, ε, ίσως δεν να σας τα πει καλύτερα η συνάδελφος Μανφρέλια. Πάντως, εν γέννη, θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ αξιόλογη η ρίσιμες και η τροπολογία. Θεωρούμε ότι λοιπόν στις προσπαθειές μας μας δίνει κίνητρο να συνεχίσουμε. Ξέρετε, χθε είχε σέντηση κορυφή για τους καταναλωτές και για την εφαρμογή του δικαίου. Γιατί θεωρούμε ότι η εφαρμογή του δικαίου είναι πυλώνας, είναι ένας βασικός άξονας για τη νέα ατζέντα του καταναλωτή είχαμε σε αυτή τη συνάντηση 450 που μέρο. μέρος ε, επίτροποι, υπουργοί. Ήρθε και η κυρία Γκέπχαρτ και άλλοι βουλευτέ. Οπότε είδαμε πώς όλοι οι εμπλεκόμενοι και όλα τα θεσμικά όργανα ενδιαφέρονται. Κύριε Μανφρέντε, έχετε το λόγο, λέει πρώτος. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Για να επανέλθω σε αυτά που είπε ο συνάδελφος Ίσως και ευκαιρία θα ήταν, αλλά βεβαίως το Κοινοβούλιο θα αποφασίσει αν θα δραχτεί της ευκαιρία αυτή να ασχοληθούμε λίγο με το κεντρικό θέμα της θεσινής ημέρας στην διάσκεψη κορυφή των ε, καταναλωτών, Consumer Summit, όσον αφορά τον χαρακτήρα της, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα είδατε ίσως ότι πολλή συζήτηση γίνεται αυτές τις μέρες ε, για το τι μπορούμε να κάνουμε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 όσον αφορά περιπτώσεις όπως το Απλουάν ας πούμε, το που ξεπερνούν ε, την αντιμετώπιση που έχουν οι παρόντες ε, κανονισμοί για τις διαστηνεριακές ε, ε, Υπάρχουν εκατοντάδες, βλέπε χιλιάδες αν όχι εκατομμύρια καταναλωτές οι οποίοι έχουν πρόσβαση ταυτόχρονα στις ίδιες υπηρεσίες. Δεν έχουμε ακόμα συγκεκριμένα πράγματα τα οποία στα οποία να έχουμε καταλήξει μετά από τις ε, συζητήσεις των δύο τελευταίων ημερών. Αλλά όλοι οι συνέλφοι της ΑΝΚΟ θα σας επιβεβαιώσουν ότι υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον ε, παρεμβάσεις και σε υπουργικό επίπεδο ε, για ε, τέτοια ε, προγράμματα και ενδεχομένως τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να επικυροποιήσουμε τον κανονισμό CPC. Η ψηφιακή ενιαία αγορά είναι σημαντική και για μας και ό,τι μπορείτε να, όσο μπορείτε να συμβάλλετε κατά αυτή την έννοια είναι καλοδεχούμενο. Το σημαντικό είναι να έχουμε μια καλή επαφή Επίσης ε, ε, θα ήθελα και εγώ όπως και ο συνάδελφός μου να καταλάβω καλύτερα την έννοια του collective consumption, συνολική κατανάλωση, συλλογική συγγνώμη κατανάλωση. Ευχαριστώ πολύ για αυτά που μας είπατε. Ο εισηγήτης τώρα. Και πάλι για να μας πήγε για το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ίσως. Ευχαριστώ πολύ. Άκουσα με μεγάλη προσοχή τις ε, απόψεις που εξετέθησαν και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν μπορώ παρά να χαρώ για την υποστήριξη που προσφέρατε. Επρόκειται εδώ για συνεργασία στην οποία βασιζόμαστε, οπότε τα συνεργασία απευθύνονται σε όλους. Νομίζω ότι προχωρούμε και προχωρούμε αξιόλογα και γι' αυτό θα πρέπει να, να δούμε ότι η ατζέντα για τον Ευρωπαίο καταναλωτή μας οδηγεί στην προοπτική της προστασίας των συμφωνών του καταναλωτή. Βεβαίω σίγουρα όλες αυτές οι προσπάθειες είναι απαραίτητες, ούτως ώστε να έχουμε την ε, εφαρμογή και την υλοποίηση αυτών των δικαιωμάτων και αυτό να γίνεται παντού στην κοινωνία από πλευράς των, ε, των ε, επιχειρήσεων και αντίστοιχα πρέπει να σας αναφέρω ότι οι τροπολογίες ε, στις οποίες κατέληξε η Επιτροπή των Μεταφορών έλεγχθη υπόψη από τις ε, συμβαστικέ τροπολογίες ε, για την προστασία του καταναλωτή και στον τομέα των ε, μεταφορών. Είναι θέμα προτεραιότητας, υψίστης. Και αυτό προκύπτει και από την τοποθέτηση της ευρωπαϊκή Επιτροπής και το έχουμε καλύψει στις τροπολογίες. Τώρα, για αυτή τη συλλογική κατανάλωση ε, είναι κάτι που θα πρέπει να μας κάνει να ψάξουμε περισσότερο το θέμα. Κάντε το έκανα και εγώ γιατί έχουμε διάφορους ε, φορείς των καταναλωτών όπου υπό την σημερινή συγκυρία είναι πλατφόρμα ανταλλαγής της κατανάλωσης με μορφές μη παραδοσιακές για προϊόντα, αγαθά και υπηρεσίες. Και μορφής συνεργατικής είναι αυτή η κατανάλωση, αυτές οι ανταλλαγές. Οπότε πρόκειται για κάποια πραγματικότητα που πρέπει να την καλύψουμε από τη νέα ατζέντα. Ισχύει οπωσδήποτε κάτι τέτοιο. Τώρα, θα πρέπει να σας επισημάνω ότι οι διασυνοριακές συναλλαγές είναι πολύ σημαντικές. Και έχουμε επίσης νέες τεχνολογίες που μας επιτρέπουν να προβάλλουμε τέτοιες συναλλαγές με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Και αυτό θα πρέπει να καλυφθεί από την νέα ατζέντα του καταναλωτή. Και τώρα και στο μέλλον. Για τα σας αναφέρω ότι έχουμε χρόνο για να καλύψουμε αυτές, αυτές τις διευκρινήσεις που έγιναν ή στο δεύτερο διάγραμμα, για να δεν κάνω λάθος. Είπαμε ότι πάμε για τις 25 Απριλίου. Οπότε και θα ψηφίσουμε στην, Ευρωπαϊκή, στην Επιτροπή μας συγγνώμη, αυτές τις συμβαστικές τροπολογίες. Στη συνέχεια δε, το Μάιο πρωτοθεώς θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε στην Επιτροπή. το σύνολο της εκθέσης. Τέλος, αυτοί οι βασικοί άξονες γύρω από τους οποίους περιστρέφονται οι σημαντικές τροπολογίες αποτελούν συνέχεια της εισήγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συζητήθηκε στο Κοινοβουλίο της Επιτροπής, οπότε και εμείς μπορέσαμε έτσι να βελτιώσουμε την πρόταση της Επιτροπής και επιτελώντας τον ρόλο που πρέπει να έχει το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Προχωρούμε στο επόμενο σημείο τα σημεία που είναι παρόμοια, το ίδιο θέμα. Προτείνω να μας παρουσιάσει σε περίπου ένα τέταρτο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων και μετά να ακολουθήσει η ανταλλαγή απόψεων με τους βουλευτές. Ε, η κυρία Ζαμπίνε Λικρινιέ είναι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε που μας προσκαλέσατε για να παρουσιάσουμε την πρόταση αναθεώρησης του κανονισμού για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα έχουμε τρεις οδηγίες, μία γενική και δύο άλλες εξειδικευμένες. Μία η οποία αφορά ε, τα ε, ειδικά ε, προϊόντα τα οποία μπορούν να εμφυτευθούν και τα άλλα τα οποία αφορούν την ε, in vitro, τα in vitro διαγνωστικά μηχανήματα. Ε, βεβαίως κύριος στόχος είναι το υψηλό επίπεδο προστασίας και των ε, χρηστών, δηλαδή αυτών που χειρίζονται τα μηχανήματα, αλλά και των ασθενών και επίσης την ελεύθερη κυκλοφορία όλων αυτών των προϊόντων με την προϋπόθεση ότι είναι ασφαλή. Στα πλαίσια ε, ε, αυτής, αυτού του ε, κανονιστικού πλαισίου θεωρούμε ότι τα κυριότερα προτερήματά του είναι η ευελιξία, είναι ο σωστός λόγος κόστους ωφέλους, η φιλικότητα προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η στήριξη της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας. Αναθεωρήσαμε το παρόν πλαίσιο πρώτα απ' όλα γιατί πρόκειται για έναν κλάδο όπου οι τεχνολογίες προωθούνται και προοδεύουν γρήγορα γρήγορα και έπρεπε λοιπόν να προσαρμοστούμε σε αυτήν την πρόοδο. Επίσης, ε, διότι διαπιστώθησαν κάποιε αδυναμίε στη λειτουργία του συστήματο ε, που έθεσαν ε, σε κίνδυνο του χρήστε αλλά και τους ασθενεί. Επίση, θελήσαμε να έχουμε διαφάνεια στην όλη διαδικασία και ίδια... Ε, αντιμετώπιση. Επίσης, ε, για να έχουμε σωστή και ομοιόμορφη εφαρμογή των ε, κανόνων και να αντιμετωπίσουμε θετικά τις προσδοκίες του κόσμου. Το Σεπτέμβριο του 12 λοιπόν, κάναμε μια ανακοίνωση για όλα τα θεσμικά όργανα, Κοινοβούλιο, Συμβούλιο, ΕΟ και, και Επιτροπή Περιφερειών και αυτή τη στιγμή έχουμε δύο προτάσεις ε, κανονισμού και όπως ε, κάθε αντίστοιχη νομοθετική ε, πρόταση, αυτές οι προτάσεις συνοδεύονται από ανάλυση επιπτώσεων, μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων δηλαδή. Ε, οι οποίες ε, καταλήγουν σε κάποιες προτάσεις και σε κάποιες ε, λύσεις. Οι διάφορες λύσεις αυτές συγκρίθηκαν και ορισμένες πήραν την τελική μορφή τους βάσει και της πολιτικής συμφωνίας. Βρίσκονται δε δημοσιευμένες στον ιστότοπό μας σε όλες τις χώρες. μετά από δύο δημόσιες διαβουλεύσεις και πολλές επαφές με τα ενδιαφερόμενα μέρη κατέληξε η μελέτη επιπτώσεων ε, σε, ορισμένες, ε, σε ορισμένα, στην ταυτοποίηση ορισμένων προβλημάτων. Ε, πρώτα απ' όλα ελλειπής έλεγχος των προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά, ε, κυρίως όσον αφορά την εποπτεία της αγοράς. Επίσης, το καταστατικό ή το, το νομικό καθεστώς των προϊόντων δημιουργεί προβλήματα. Έλλειψη χνηλασιμότητας και διαφάνειας διαπιστώθηκε, καθώς επίσης και ελλείψεις ε, όσον αφορά την προσφυγή σε εξωτερική πραγματογνωμοσύνη ε, και ελλείψεις επίσης όσον αφορά τον σαφή καθορισμό των υποχρεώσεων όλων των εμπλεκόμενων οικονομικών φορέων. Επίσης ε, και κάποιες αδυναμίες οι οποίες σημειώθηκαν στο ίδιο το κανονιστικό πλαίσιο. Αναλύθηκαν λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία έτσι ώστε ε, να ληφθούν ε, μέτρα ε, για να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας για την ανθρώπινη υγεία και για την ασφάλεια, για την διασφάλιση της καλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και έτσι ώστε να υπάρξει ένα κανονιστικό πλαίσιο το οποίο θα στηρίζει την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα. Επίσης, λήφθησαν και συγκεκριμένα μέτρα έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τα επιμέρους προβλήματα τα οποία προηγουμένως ανέφερα τα κοινά προβλήματα ε, για όλα τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τα οποία ανέφερα προηγουμένως, ε, είναι συστημικά και αντιμετωπίζονται στο πρώτο ε, τμήμα της μελέτης εκτίμησης επιπτώσεων. Πέρα από αυτό όμως υπάρχουν και δύο εξειδικευμένα κεφάλαια τα οποία αφορούν προβλήματα, τα οποία αφορούν είτε τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα εκτός των διαγνωστικών προϊόντων και τα εξειδικευμένα προβλήματα των ε, διαγνωστικών ε, ιατροχειρουργικών προϊόντων. Ε, έχουμε διαπιστώσει και στις δύο περιπτώσεις ελλείψεις όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, ανάγκη προσαρμογής σε κανονιστικές εξελίξεις, τεχνολογικές εξελίξεις και βεβαίως ανάγκη ανάπτυξης περισσότερων κλινικών δοκιμών. Ε, όσον αφορά τις, τα in vitro διαγωνιστικά προϊόντα και εδώ διαπιστώσαμε προβλήματα όσον αφορά το εύρος ε, της ε, οδηγίας, κάποιες ασάφειες και κάποιες ελλείψεις ρυθμιστικές, κάποιο προβλήμα όσον αφορά την ταξινόμηση των in vitro διαγνωστικών προϊόντων και οπωσδήποτε ανάγκη προσαρμογής σε τεχνολογικά, στις τεχνολογικές εξελίξεις, επιστημονικές κλπ. Ε, έχουν καθοριστεί και οι επιλεγήσεις ε, ε, οδοί προς την επίλυση των προβλημάτων πρέπει να πω ότι μετά την ολοκλήρωση της μελέτης εκτίμησης επιπτώσεων έλαβαν χώρα ε, τα ε, γνωστά προβλήματα τα οποία γνωρίζετε. Μετά από, την, ε, μετά από τις δοκιμές ΠΙΠ οδηγηθήκαμε σε κάποια μέτρα τα οποία θα μας επέτρεπαν να ταυτοποιήσουμε πιο γρήγορα τέτοιου είδους καταστάσεις και περιπτώσεις. Ε, είδαμε ότι οι προτάσεις ήταν σωστές, αλλά ε, ότι παρόλα αυτά έπρεπε να προσθεθούν και κάποια στοιχεία, κυρίως όσον αφορά την λειτουργία ε, των οργάνων κοινοποίησης, όσον αφορά την ταυτότητα των εμφυτευμάτων και όσον αφορά τον καθορισμό ενός ατόμου υπευθύνου για τις ρυθμιστικές επιπλοκές, όπως ακριβώς προέκυψε και στην προκείμενη περίπτωση. Να προχωρήσουμε σχηματικά στις κύριες ε, τροποποιήσεις που προτείνονται, τις οποίες μπορούμε να ομαδοποιήσουμε σε πέντε ε, στοιχεία. Πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, ε, υποχρεώσεις πριν από την θέση στην αγορά, κυκλοφορία στην αγορά, καθώς και υποχρεώσεις μετά την κυκλοφορία στην αγορά, η διαφάνεια και η διακυβέρνηση του συστήματος. Πρώτα απ' όλα, πεδίο εφαρμογής. Το πεδίο εφαρμογής των οδηγιών διευρύνθηκε. Προτείνεται ε, να καλύπτονται τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ε, τα οποία χρησιμοποιούν ε, είτε ιστούς είτε κύτταρα μη βιώσιμα. Επίσης, ε, αποφασίστηκε ότι οι ε, ας πούμε αισθητικές παρεμβάσεις ε, οι οποίες χρησιμοποιούν προϊόντα τέτοια αφομοιώνονται πλέον, εξισούνται με τις αντίστοιχες που έχουν ιατρικό σκοπό. Επίσης αποφάσεις ελήφθησαν όσον αφορά την ανακύκλωση των προϊόντων μιας χρήσης Επίσης ε, τα γενετικά τεστ, οι γενετικές ε, δοκιμές ε, οι οποίες ταυτοποιούν την προδιάθεση για κάποια ασθένεια ή για κάποια περιπλοκή ε, επίσης ε, όλες αυτές τις συνοδευτικές διαγνωστικές ε, μελέτες και έρευνες οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στην καλύτερη αντιμετώπιση του ασθενούς. Επίσης ότι οι δοκιμές in-house θα πρέπει να γίνονται λαμβάνοντας υπόψη τους σχετικούς κινδύνους. Επίσης εδώ στο πεδίο συμπεριλαμβάνονται πλέον και οι συσκευές οι οποίες χρησιμοποιούνται για εξαποστάσεως διαγνώσεις. Ε, όσον αφορά τώρα την ε, ε, ε, ταξινόμηση κινδύνου πριν μπουν τα προϊόντα στην αγορά. πρώτα απ' όλα έχουμε καλύτερη, έχουμε λάβει περισσότερο υπόψη και την εμπειρία εφαρμογής των ε, παρόντων κανόνων και τις τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις ε, και όλα τα ε, νέα στοιχεία. Πρέπει να σας πω ότι έχουν αλλάξει πλέον πολύ και οι συνθήκες όσον αφορά τα in vitro διαγνωστικά προϊόντα. Πλέον βρισκόμαστε σε ένα νέο σύστημα με λογική τάξεων από την α μέχρι την δ. Ε, μέχρι τώρα στοιχεία και προϊόντα τα οποία ε, ήλεγχε μονάχα ο κατασκευαστής πλέον ελέγχονται από ε, συγκεκριμένους φορείς. Όσον αφορά τώρα τα σώματα κοινοποίηση, είναι πιο αυστηροί και πιο λεπτομερείς οι ε, κανόνες ελάχιστων νομικών απαιτήσεων. Έχουμε ε, ενιαία πρακτική όσον αφορά τον καθορισμό και την εποπτεία ε, και βεβαίως έχουμε πλέον κοινή αξιολόγηση με εκπροσώπους και της Κομισιόν και των κρατών μελών. Επίσης έχουν ενισχυθεί τα σώματα αυτά μέσα από ξαφνικές ε, επισκέψεις ε, στους ε, κατασκευαστές μέσω περιτροπής των, του προσωπικού καθώς επίσης και ενός μηχανισμού ελέγχου κυρίως για τις συσκευές και τα προϊόντα υψηλού κινδύνου. Προτείνονται επίσης βελτιώσεις όσον αφορά τα, τις, τα κλινικά ευρήματα ε, με καλύτερη αξιολόγηση των κλινικών δεδομένων που πρέπει να υποβάλλονται πριν την ε, κυκλοφορία στην αγορά, αλλά και με υποχρέωση παροχή στοιχείων follow-up ε, μετά βάση των κλινικών στοιχείων που παρουσιάζονται στην αγορά μετά την ε, ε, διεμπόρευση ε, έχουν προσθεθεί και ενισχυθεί μέτρα εποπτείας και ελέγχου της αγοράς, κεντρική διαδικασία αναφοράς των σοβαρών περιπτώσεων, καλύτερος και εντονότερος συντονισμός μεταξύ των εθνικών σημείων επαφής, ανάλυση τάσεων καθώς επίσης και μέτρα που αφορούν το σύνολο της ε, ε, ε, διαδικασίας. Ένα σημαντικό σημείο στην αναθεώρηση ήταν η διαφάνεια. Βελτιώνουμε τη διαφάνεια μέσα από ένα κεντρικό σύστημα καταχώρησης και των operators και των προϊόντων. Έχουμε επίσης προβλέψει μία περίληψη των χαρακτηριστικών κλινικών επιδόσεων και ασφάλειας. Έχουμε πλέον και ένα καινούριο καινούριο σύστημα ιχνηλασιμότητας βάσει ε, μιας ε, ε, ενιαίας και μοναδικής συσκευής ταυτοποίησης και έχουμε και μια implant card για κάθε προϊόν. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο αντιμετωπίσαμε ήταν το θέμα της διακυβέρνησης. Οι προτάσεις μας δημιουργούν ένα νέο σώμα ε, συντονισμού των ιατρικοτεχνολογικών ε, προϊόντων με συγκεκριμένη τεχνική, επιστημονική και ε, λογιστική στήριξη από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, ε, προβλέπεται και διαρθρωμένη επικοινωνία μεταξύ ε, των ε, εξωτερικών εμπειρογνωμόνων μέσα από τη δημιουργία κάποιων εργαστηρίων της, που θα αποτελέσουν αναφορά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τώρα περνάμε στη συγγήτρια. Α, η κυρία Μπέρα. Σας βλέπω, ναι. Την είδα την κυρία Μπέρα. Euh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρώτα-πρώτα θα πρέπει να ευχαριστήσουμε ε, την Επιτροπή που εξεπώνησε αυτό το κείμενο η οποία ε, έτσι ε, ανέδειξε όλα αυτά τα προβλήματα όσον αφορά αυτό το, το ιατρικό υλικό ε, και εσείς, ε, αυτά τα ιατρικά προϊόντα τέλο πάντων σε σχέση με την εποπτεία, με τον έλεγχο της αγοράς, ούτως ώστε να φτάσουμε σε κάποια εναρμόνιση των θεσμοθετημένων υποχρεώσεων. Και οπότε, όπως είπαμε, θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα σκάνδαλα τα οποία έχουν πάρα πολύ υπονομεύσει την ε, εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων. οπότε και γι' αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει. Γιατί έχουμε βέβαια στις Ηνωμένε Πολιτείε μόνο έναν φορέα για αυτά τα προϊόντα, τα ιατροτεχνολογικά. Ενώ εδώ στην Ευρώπη έχουμε 80 προϊόντα πιστοποίηση. Ε, ούτως ώστε να μπορέσει στις 27 διαφορετικές χώρες να κυκλοφορήσει το ίδιο προϊόν. Άρα θα πρέπει να πασχίσουμε ούτως ώστε να εξεύρουμε μια εγγύηση ομοιομορφίας των ελέγχων ομοιομορφία στην ε, ασφάλεια αλλά και την ποιότητα των προϊόντων που κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά. Επομένως, με αυτόν τον ε, ε, κανονισμό, κωδικοποιούνται όλα, όλες οι φάσεις στην ζωή, στην πορεία της προϊόντος, ε, πριν και μετά τη θέση σε εμπορία για τους πιστοποιημένους οργανισμούς που εποπτεύουν επομένω όλη την πορεία πριν και μετά τη θέση σε εμπορία. Οπότε για να δούμε τώρα στον αφορά το πεδίο εφαρμογή του κανονισμού. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε διάφορα προϊόντα που ονομάζονται αισθητικά, τα οποία ε, έχουν παρόμοιο χαρακτήρα με τα ιατροτεχνολογικά, τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πρόβλημα στη δημοσιογή. Έχουν καλυφθεί από το κείμενο παρόλα αυτά. Εδώ το ότι τα βάζουμε στον ορισμό για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα έρχεται σε σύγκρουση ε, με, με, με, την, με τον βασικό χαρακτηρισμό αυτών των προϊόντων, δηλαδή τον ιατρικό τους χαρακτήρα. Επίσης, στο, και στο παράρτημα έχουμε πρόβλημα που όλα αυτά τα προϊόντα που μπαίνουν εκεί δείχνουν τη δυσκολία της προσαρμογής και επικαιροποίηση που θα πρέπει να γίνει οπότε θα πρέπει να δούμε κατά πόσο έχει αποκλειστικό χαρακτήρα και ε, εξαντλικό αυτή η, η λίστα, αυτός ο κατάλογος. Ε, οπότε για όλα αυτά τα αισθητικά και μη ιατρικά προϊόντα ε, θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη να κρυφθούμε από τον κανονισμό. Όσον αφορά τώρα τις υποχρεώσεις των ε, οικονομικών συναλλασσομένων, εδώ καλύπτονται όσον αφορά την υποπτία για την ποιότητα των προϊόντων, για την εποπτεία μετά τη θέση εμπορία και κατόμενη των σχετικών σκανδάλων είναι απαραίτητο να κατοχυρωθεί ο ασθενής κατά του ε, κατασκευαστεί σε περίπτωση υπέρευσης κάποια ζημία. Το θέμα είναι τώρα πώς θα έχουμε εγγύσεις, ούτως ώστε να υπάρχει αποζημίωση πλήρης σε περίπτωση που κάποιος ασθενής επομένως υποστεί κάποια βλάβη. Ίσως μπορούμε εδώ πέρα να εντάξουμε μια ε, διάταξη, κάποια ρήτρα που συνδέεται με μια ασφάλεια, μια ασφάλιση. Πρέπει να μας προβληματίσει αυτό. Επίσης τώρα το θέμα των ευθυνών που έχουν οι, <clears throat> οι operators ε, σε σχέση με τα προϊόντα αυτά. Χρειάζεται κάποια επαγρύπνηση που προβλέπει ότι ένας ε, εισαγωγία θα πρέπει να λαμβάνει διορθωτικά μέτρα αν χρειάζεται στο βαθμό που μπορεί να έχουμε όμως περισσότερους ε, εισαγωγείς πρέπει να έχουμε και περισσότερα διορθωτικά βήματα και αυτό να γίνεται αποκλειστικά για όχι για, το, για, τον, για τον κατασκευαστή, αλλά για να έχουμε συνοχή, αυτό να το κάνουν μόνο οι εισαγωγές ή ο εισαγωγές. Για την ανακύκλωση του τρότου μιας χρήσης, θα πρέπει και αυτό να καλυφθεί ε, στο άρθρο 15. Ίσως θα, θα πρέπει να επισημαίνεται στον κατασκευαστή. Ορισμένοι λένε ότι για λόγους εμπορικούς ε, γίνεται κατάχρηση της δυνατότητας που έχει ο κατασκευαστής. Άρα θα πρέπει να γίνει μια αυστηρή ρύθμιση σχετικά με αυτό το τρόπο αφορά για τα ε, προϊόντα τα οποία αποσκοπούν στη χρήση σε περιπτώσεις ανάγκης και εδώ θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση από τις, πιο, τις τελευταίες επιστημονικές ανακαλύψεις. Γιατί εδώ πέρα είναι πολύ αόριστη διατύπωση. Επίσης, προς την Κομισιόν θα πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε κάποιες κοινέ ε, ε, ρυθμίσεις. Πώς θα... Πώς, πώς θα, η επάρκεια των ε, κανόνων που προβλέπονται Πώ θα κρυθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, όσον αφορά του κοινωνικού οργανισμού, έχουμε σήμερα ε, πρόβλημα το ότι ένα κατασκευαστή ελεύθερα μπορεί να διαλέξει τον οργανισμό επιστοποίηση. όποιον θέλει από τους 18 που συνεπάρχουν στην Ευρώπη. 18, 18. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτή η ελευθερία του ε, επιτρέπει να έχουν μια σχέση εμπιστοσύνη. Ε, και επομένω εδώ πέρα είναι θέμα αντικειμενικότητα και ποιότητα των ελέγχων που ελέγχονται επίση. Ε, όμως ε, είναι αόριστη η σχέση και το όριο μεταξύ συμβουλής και πιστοποίησης. Ε, θα πρέπει να υπάρχει πιστοποίηση και για, τα προϊόντα που ενέχουν κινδύνους, θα πρέπει να γίνεται κλινική αξιολόγηση. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό οι κοινοποιημένοι οργανισμοί που κάνουν αυτή την αξιολόγηση για τα ευαίσθητα προϊόντα να έχουν εμπειρογνωμοσύνη όπως απαιτείται. Οπότε στο μέτρο του δυνατού αυτή η εμπειρογνωμοσύνη να, να, να, να, να, να κρίνεται αν δεν θέλουμε σύγκρουση συμφέροντων. Γίνονται βήματα πρώτα επομένω, αλλά χρειάζεται να βελτιωθεί το κείμενο. Όσον αφορά τώρα την κατηγοριοποίηση, την κατάταξη, θα πρέπει Ε, να δούμε ε, το πώς θα πάνε τα προϊόντα τα οποία λαμβάνουν το στόμα ή οι σπνέοντες να μπουν στην τρίτη κατηγορία. Και να δούμε τι θα γίνει με τα προϊόντα που θεωρούνται οριακά, borderline. Τα αντιόξινα, όλα αυτά θα πρέπει να χαρακτηριστούν ανάλογα με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που σχετίζονται με αυτές τις ουσίες. αυτά τα οποία τα λοιπόν συστηματικά θεωρούνται φάρμακα. Να πάνε στην τρίτη κατηγορία και να θεωρηθούν ιατρικά προϊόντα. Κατηγορούμε εδώ μπαίνουν πάρα πολλά γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να κατατάξουμε 6.000 προϊόντα δύσκολο να τεθούν επομένω οι κανόνε τη ε, κατάταξη εάν δεν περάσουν από κάποια επεξεργασία. Όσον αφορά την αξιολόγηση τη συμβατότητα, είναι από τα πιο προβληματικά σημεία του κειμένου, όπως είπαμε, εδώ πέρα υπάρχει πραγματικά πρόβλημα τη ε, ενιαία αντιμετώπιση. γιατί οι ενεργητικοί μηχανισμοί, όπω προβλέπονται από το άρθρο 44, με τον συντονισμό αυτών των ε, προϊόντων, έχουμε τώρα αυτό το δικαίωμα ελέγχου από πλευράς της διάταξης που τελικά δεν βοηθάει κανένα για κάποιες ε, αρχές γεωνομικές, για τους ε, ασθενείς, τους καταναλωτές. Δεν έχει αρκετά δεσμευτικό χαρακτήρα αυτό το άρθρο. Γιατί χρειάζεται να γίνει πιστοποίηση, να συμπληρωθεί η πιστοποίηση. Άρα για την έρευνα ε, αυτό είναι μια δυνατότητα και έχει μια υποχρέωση. Θα πρέπει να υπάρχει όσο καθώς ορισμός. Θα πρέπει να αποφασίζει η ομάδα συντονισμού με απλή πλειοψηφία και ακόμα και αν δεν έχω έχουν και αποφάσει αυτού του οργάνου, μια αρνητική γνωμοδότηση θα επηρεάζει τη θέση σε εμπορία του Τώρα θα δούμε τι θα γίνει μετά με τι ΜΜΕ, τα έξοδα τη καινοτομία και πότε θα πρέπει και αυτό θα πρέπει να δούμε πώς θα είναι η προσέγγιση ρεαλιστική. Ναι, ναι, ναι, θα, θα τελειώσω τώρα, Πρόεδρε. Δύο λεπτά, δύο λεπτάκια. Θα πρέπει επομένω να ανταποκριθούμε σε αυτό το οποίο θέλουν οι ασθενεί, δηλαδή ε, έναν έλεγχο ε, από το δημόσιο, κρατικό έλεγχο, ούτω ώστε να μπορούμε με αποτελεσματικό τρόπο να διατηρήσουμε το ισχύον σήμερα πρότυπο. Όσον αφορά την κλινική αξιολόγηση, να σα πω δύο λόγια, γιατί η ισχύουσα νομοθεσία δεν εφαρμόζεται ορθά οι έρευνες είναι, είναι δυνατόν να, να, να μην ισχύσουν εάν αποδείξει το ότι ο αποδείξει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος και να υπάρχει ισοδύναμη διάταξη. Επομένως, θα πρέπει να καταλήξουμε στο ότι το σχέδιο ο ε, κανονισμού αυτού θα πρέπει να καλύψει και τα implants στην τρίτη κατηγορία. Οπότε ε, είναι και, ε, πρέπει να δούμε τι θα γίνει, πώς, με ποια μεθοδολογία θα γίνει η αξιολόγηση και με ποιο στόχο θα γίνει η αξιολόγηση. Χρειάζεται υποπτία και μετά τη θέση εμπορία αυτών των προϊόντων Διακόπτη πρόεδρο. Ναι, ναι, τελειώνω, τελειώνω. Οπότε, απλώ να σας πω όσον αφορά την επαγρύπνηση στην αγορά, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και καινοτόμο βήμα. Τα προϊόντα που αφορούν τη διάγνωση είναι σημείο στο οποίο δεν, δεν μπόρεσα να, να, να ερευνήσω και για τα, για τα προϊόντα επομένω in vitro, τα διαγνωστικά. Κάντε ένα διάλειμμα πρώτα αν έχετε την καλοσύνη. Πρώτον, γιατί ζητούν πολλοί συνάδελφοι το λόγο και δεύτερον, αφού υποβληθεί η εκθεσή σας, θα έχουμε τουλάχιστον δυο φορές ακόμα την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτό το σημαντικό, καυτό θα έλεγα θέμα, για να το συζητήσουμε στην Επιτροπή να ακούσουμε τους άλλους σκιώδεις και τους συναδέλφους που ζήτησαν το λόγο. Ο συνάδελφος από τους σοσιαλδημοκράτες και σοσιαλιστές. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν να συγχαρώ την συνάδελφο εισηγήτρια που υπέβαλε πλήρη ανάλυση, ολοκληρωμένη πρόταση νομοθετική. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν την ώρα μπέρα. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πολύ αποτελεσματική ενημέρωση της εξηγήσει. Τα σχόλιά μου, πρέπει να σας πω, δεν αφορούν μόνο αυτή την πρόταση νομοθετικού περιεχομένου, αλλά θα καλύψουν και τις διατάξεις για τα in vitro προϊόντα, που είναι συναφή για να μην επαναλαμβάνω τα ίδια όταν μιλήσουμε για την άλλη έκθεση. Είχαμε ένα πρόσφατο σκάνδαλο το οποίο το πρόσεξαν όλοι. Αυτό αναφέρθηκε και στο New England Journal of Medicine τον Ιανουάριο και αφορούσε τις διαφορές μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένε Πολιτείε σχετικά με το, τους ρυθμιστικούς φορείς. Αναφέρθηκαν αυτά και από τη συνάδελφα Ροτ Μπέραντ. Κάνουμε εδώ μια σύγκριση των ρυθμιστικών φορέων για τα προϊόντα αυτά. Τα προϊόντα τα βλέπουμε καμιά φορά ως παρόμοια, ενώ στην πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετικά. Και επειδή είμαστε μια κοινότητα 27 κρατών μελών, ε, διαφέρουμε σε αυτό το στάδιο από τις Ηνωμένε Πολιτείες τώρα τουλάχιστον. Επίσης να έχουμε υπόψη μας ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με φαρμακευτικά προϊόντα. Θα χρειαστεί λοιπόν εθνική πραγματογνωμοσύνη στα κράτη-μέλη και εδώ υπάρχουν δυναμίες. είναι δύσκολο να υπάρχει ένας δημόσιος φορέας που θα ασκεί αποτελεσματική ρυθμιστική λειτουργία εδώ. Αυτό όμως χρειάζεται. Στη χώρα μου το σύστημα είναι δημόσιο, αλλά είναι αναποτελεσματικό. Καλύτερα θα ήταν να έχουμε μια άλλη ρύθμιση μαζί που θα συνεργάζονται με τους κοινοποιημένους οργανισμούς. Τώρα για την έγκριση, για την εμπορία. Υπάρχουν ε, προβλέψεις, αλλά δεν νομίζω ότι η έγκριση θα πρέπει να είναι υπερβολική, να είμαστε απαιτητικοί, αλλά όχι υπερβολικοί. Γιατί δεν θέλουμε το μηχανισμό αυτόν να τον χρησιμοποιήσουμε για να αναθεωρήσουμε όλα τα προϊόντα. Τα περισσότερα καλύπτονται από τις κατηγορίες 1 και 2β, οπότε δεν χρειάζεται εμείς να ε, πιέσουμε την κατάσταση και να κάνουμε υπερρύθμιση περισσότερο από ό,τι χρειάζεται. Συμφωνώ με τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η μεγάλη επένδυση που πρέπει να γίνει θα πρέπει να γίνει στη φάση μετά την εμπορία, μετά την κυκλοφορία. Χρειαζόμαστε μηχανισμούς ιδιαίτερα αυστηρούς και τα συστήματα ενημέρωσης πρέπει να είναι απόλυτα λειτουργικά. Θα πρέπει να υπάρχει ομαλή ροή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό είναι ο καλύτερος μηχανισμός και να υπάρχει καταχώρηση. Δεν μπορεί να έχουμε κλινικές δοκιμές όπως ε, γίνονται στα φάρμακα, σε αυτά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Ούτε έχουμε τόσο υψηλής ε, αξιοπιστίας ε, βάσης δεδομένων για αυτά τα τελευταία. Θα είναι δύσκολο λοιπόν να γίνουν. Πολλές φορές είναι δυνατόν να γίνουν και κλινικές δοκιμές. Όποτε είναι δυνατόν να γίνονται, πρέπει να γίνονται βέβαια. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο και θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση στη φάση μετά την κυκλοφορία στην αγορά για να γίνεται σωστή συλλογή πληροφοριών. Είναι δύσκολο να γίνονται συγκρίσεις βέβαια γιατί πολλές φορές η κλίμακα είναι πολύ μικρή. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία πολύ ενδιαφέροντα. Θα πρέπει να δούμε γιατί δεν προχώρησαν οι διαδικασίες ε, κατά την προηγούμενη θητεία. Θέλουμε πιο, πιο πολλά στοιχεία πολλές φορές από τους κατασκευαστές και για την ε, διακυβέρνηση ε, έχουν έναν ενιαίο φορέα στη ΣΥΠΑ, εμείς έχουμε πολλούς φορείς στα κράτη-μέλη μας. Πολλές φορές ε, είναι απρόθυμοι φορείς αυτοί να συνεργαστούν λόγω των τεχνολογικών καινοτομιών σε αυτόν τον τομέα. Αν ε, δείτε τους εθνικούς, τι γίνεται σε εθνικό επίπεδο, χρειάζεται πολλές φορές να δημιουργηθεί ένας κορμός τεχνογνωσίας. Ε, υπάρχουν διαφορές όπως είπαμε, τα φάρμακα και το πώς χειρίζεται τα φάρμακα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων. Είναι διαφορετικά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Πάντως, νομίζω ότι υπάρχουν πολλά υπέρ στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να μην έχουμε μόνο αποκεντρωμένη οργάνωση, αλλά να έχουμε παράλληλα και μια ε, συγκεντρωτική ομάδα, συγκεντρωμένη ομάδα εμπειρογνωμόνων Μπορεί ίσως κάποια στιγμή να χρειαστεί και ένας ευρωπαϊκός οργανισμός για να τα δει όλα αυτά, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το βαθμό οριμότητας για να ε, προσεγγίσουμε και να αποκτήσουμε τις πληροφορίες με αυτόν τον τρόπο. Είναι σημαντικό να έχουμε πληροφορίες για προσφορά και ζήτηση, αλλά και κατάλληλη πληροφόρηση ε, μεταξύ των ρυθμιστικών φορέων. Χρειάζεται δουλειά και στην ε, επισήμανση, στη συσκευασία για καλύτερη χνηλασιμότητα, για εντοπισμό παραποιημένων, μείωση των ανεπιθύμητων συμβάντων και βελτίωση τη ενδυνάμωση ενιαίας αγοράς. Λοιπόν, η κυρία Παρβάνοβα, εξ ονόματος των φιλελευθέρων. Θα μιλήσετε εσείς για τους φιλελευθέρους. Α. Κύριος Μάντερς. Ναι, και για την ΕΝΒΗ. Έχω μόνο μία ερώτηση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί είπαμε τη μία μεριά έχουμε το αμερικανικό σύστημα και την άλλη το ευρωπαϊκό. Και μετά από όλη αυτή την διαφήμιση, τι γίνεται, τι γίνεται με την ασφάλεια. Ποιος, ποια, ποιο σύστημα από τα δύο παρέχει περισσότερη ασφάλεια στον ασθενή. Dankeschön, Frau Rühle von den Grünen. Also ich habe mich nur gemeldet, weil ich... Εγώ ζήτησα το λόγο γιατί εντυπωσιάστηκα από τις γνώσεις της εισηγήτριας αφενός, αλλά φοβούμε αφετέρου ότι θα έχουμε εδώ μία έκθεση που οδηγεί σε επικάλυψη με την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Εμένα με ενδιαφέρει το συγκεκριμένο ποσοστό δηλαδή της, που, της ε, ενασχόλησης της δικιάς μας Επιτροπής, γιατί θέματα που κάλυψαν άλλες επιτροπές δεν πρέπει να τα καταφιαστούμε κι εμείς. Σε αυτό επιμένει η πολιτική μου ομάδα, να ε, υπάρχει σαφής οριοθέτηση, ούτως ώστε να αποφεύγονται επικαλύψεις στο έργο των Επιτροπών. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω άλλους να ζητούν το λόγο από τις άλλες ομάδες και έτσι περνούμε στους υπολείπους βουλευτές που θέλουν να ε, μιλήσουν. Ο κύριος Φόξ. Δεν ξέρω αν με έχετε στο κατάλογο, αλλά εγώ είμαι παντού σκιώδη συζητητή για του ε, συντηρητικού μεταρρυθμιστέ. Να, να, να, μια ευχάριστη έκπληξη. Εγώ είμαι. Ωραία. Είναι σειρά σα, λέει ο πρόεδρο. Πρόεδρε, θα ήθελα απλώ να σα πω ότι ε, όσον αφορά αυτά τα εμφυτεύματα PIP, υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Οπότε, η ρύθμιση και η νομοθεσία πρέπει να βελτιωθεί. Νομίζω ότι γίνονται βήματα πρόοδου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί έτσι ενδυναμώνεται οι κοινοποιημένοι οργανισμοί, υπάρχουν εναλλακτικά μέτρα. Η εναλλακτική λύση πάντως θα ήταν να έχουμε μια κεντρική ευρωπαϊκή υπηρεσία. Κάτι γνώμη μας, όμως όσον αφορά τις ε, συσκευέ, ε, δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα σύστημα πιο αργό, πιο ακριβό, όσον αφορά και θα, δεν θα, διευκολυνθεί η προσβασιμότητα. Πριν την θέση εμπορία θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος ε, των συσκευών, να ενθαρρύνονται επομένω οι υπάρχοντες οργανισμοί, να υπάρχει περισσότερη παρρύπνηση και με τη θέση εμπορία για να είναι τόσο το σύστημα λιγότερο γραφειοκρατικό. Επομένως, να γίνεται επαρρύπνηση αγοράς Καλύτερο συντονισμό και σε και από την νομοθεσία αλλά και στη φάση κατασκευαστική θα πρέπει να υπάρχει εποπτεία. Και εδώ τελειβάζουμε τελεία γιατί ξέρω ότι σε πέντε λεπτά πρέπει να είστε μετρήσουν συντονιστές. Δύο ακόμη ζητούν το λόγο, προλαβαίνουμε. Μετά σύντομα θα λάβουν το λόγο η Επιτροπή και η, η συγγήτρια. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάδελφο που παρουσίασε αυτήν την έκθεση και να ευχαριστήσω βεβαίως και την Κομισιόν για τις παρατηρήσεις. Ε, υπάρχουν κάποια βασικά προβλήματα μεταξύ των οποίων αναφέρθηκε και η χνηλασιμότητα αυτών των προϊόντων γιατί τα κράτη-μέλη του τη στιγμή δεν είναι σε θέση, δεν έχουν ε, συνολικές πληροφορίες όσον αφορά τη διανομή των προϊόντων αυτών. Μια ερώτηση προς την Κομισιόν φαίνεται ότι βομβαρδίζεται η εσωτερική αγορά από προϊόντα προέλευσης τρίτων χωρών, ασαφούς στην ουσία προελεύσεων, ε, που στην ουσία φτάνουν στην, από τρίτες χώρες ε, ε, και μέσα από τροποποίηση της συσκευασία τους προωθούνται σαν ευρωπαϊκά προϊόντα. Επομένως, ο καταναλωτής δεν μπορεί να έχει μια σωστή, να κάνει μια σωστή αξιολόγηση αξιολόγηση της κατάστασης και βεβαίως αυτά είναι προϊόντα τα οποία απευθύνονται σε μη ε, επαγγελματίες η Κομισιόν το ξέρει το πρόβλημα το συζητάει προβλέπει κάτι ο κύριος Βάπ Ευχαριστώ μια και είμαι τελευταίος θα είμαι σύντομο. Είπαμε να μιλήσουμε και για τη μελέτη εκτίμηση των επιπτώσεων ε, από την Επιτροπή. Ε, παρακλίναμε λίγο. Τώρα, για τις καταχρήσεις και τις απάτες. Εδώ δεν θα μας βοηθήσει ούτε ο νέος κανονισμός και αυτό ήταν σημαντικό ε, μετά το μεγάλο σκάνδαλο με τα ενθέματα του μαστού. Η Κομισιόν πάνω στη βάση της μελέτης επιπτώσεων θα πρέπει να κάνει βελτιώσεις και να έχουμε έναν κανονισμό ε, που θα αναγκάζει όλα τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν τους κανόνες όπως ακριβώς αναφέρονται μέσα στον κανονισμό. Και υπάρχει και μια σειρά από σημεία και ο κύριος Φόξ και η κυρία Μπέρα, η συγκήτριά μας, τα ανέφεραν που είναι σημαντικά. Πάνω από όλα η εποπτεία της αγοράς και το είπατε και εσείς σε άλλο πλαίσιο κυρία Πρόεδρε η εποπτεία της αγοράς θα πρέπει να ενισχυθεί και να υπάρχει καλύτερος έλεγχος αεφνίδι, έλεγχοι στα εργοστάσια θα πρέπει. Υπήρχαν και ε, προβλέπονταν από την παλιά οδηγία, αλλά δεν γινόντουσαν τον παλιό κανονισμό. Θα πρέπει λοιπόν να μην μας ε, εμποδίσει η γραφειοκρατία ε, να συνεχιστούν οι καινοτομίες στα ιατροτεχνολογικά και να παίρνουν οι ασθενείς καινοτόμα προϊόντα αποτελεσματικά και ασφαλή. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, η Κομισιόν Θέλετε να απαντήσετε σε κάποιες ερωτήσεις που ακούσαμε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πολύ σύντομα να απαντήσω στην ερώτηση για ε, όσον αφορά τη σύγκριση με το αμερικανικό σύστημα. Άλλες μελέτες λοιπόν καταλήγουν ε, ότι το ευρωπαϊκό σύστημα είναι καλύτερο και πιο ασφαλές, άλλες ότι το αμερικανικό είναι πιο ασφαλές από το άλλο. Πάντως σε γενικές γραμμές εγώ πιστεύω ότι είναι περίπου ίδια τα προγράμματα, αλλά το βέβαιο είναι ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα επιτρέπει, αφήνει περισσότερο χώρο για την καινοτομία, επιτρέπει πιο γρήγορη πρόσβαση των νέων νέων προϊόντων ε, στην ε, αγορά. Ε, πάντα βέβαια με τις προϋποθέσεις που ανέφερα προηγουμένως. Όσον αφορά τώρα την πρώτερη αδειοδότηση και τα λοιπά, για λόγους που σχετίζονται με την πληθώρα των προϊόντων ε, είναι κάπως βραδία η ε, επικεντρωμένη διαδικασία, αλλά βεβαίως στο άρθρο 44 προβλέπεται δυνατότητα ελέγχου ε, που αποσκοπεί αφενός ε, να ε, γνωρίζουν τα κράτη-μέλη ποια είναι τα καινοτόμα προϊόντα που φτάνουν στην αγορά και αφετέρου ε, να ελέγχονται σε ορισμένες περιπτώσεις οι οργανισμοί πιστοποίησης καθώς επίσης να υπάρχει και δυνατότητα συγκρίσεων των κλινικών αποτελεσμάτων στα οποία έχουν καταλήξει ή επί των οποίων έχουν βασιστεί αυτοί οι οργανισμοί πιστοποίησης και τέλος έτσι ώστε να γίνουν σεβαστές ε, σεβαστεί κάποιοι κανόνες οι οποίοι διέπουν ε, συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, πράγμα που λείπει από τον σημερινό κανονισμό. Όσον αφορά τώρα τις ευνηδιαστικές επισκέψεις ε, και τους ελέγχους χωρίς προειδοποίηση, βεβαίως είναι ένα από τα μαθήματα που μάθαμε από το θέμα των εμφυτευμάτων μαστού PIP να γίνονται οι έλεγχοι όχι μονάχα άλλωστε στο τόπο κατασκευή, στο εργοστάσιο, αλλά ε, και στην αγορά, στους τόπους χρήσης, σε συνοδεία και των εθνικών αρχών που θα πρέπει ε, στην, στα πλαίσια της εποπτείας της αγοράς να παίρνουν και δοκίμια. Πράγμα που δεν ε, έγινε στην περίπτωση των εμφυτευμάτων PIP. Επίσης, ε, όσον αφορά την ιχνηλασιμότητα, σιγά σιγά και ξεκινώντας από τα προϊόντα υψηλότερου κινδύνου, θα εφαρμόσουμε, λέω, ένα σύστημα ε, ιχνηλασιμότητας, έτσι ώστε να μπορούμε να ξεκινήσουμε από τον χώρο ε, κατασκευής στην Ευρώπη σε μια τρίτη χώρα και μετά να καταλήγουμε στην άλλη άκρη, στο νοσοκομείο ή στον μεμονωμένο ασθενή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και στο τέλος η εισηγήτρια. Και σας ερωτώ, το θέμα είναι τόσο καυτό στην κοινή γνώμη και το μεγάλο ενδιαφέρον και στο Κοινοβούλιο επίση δείχνει πόσο σημαντικό έχει γίνει το θέμα. Ίσως θα πρέπει να διοργανωθεί μια ακρόαση ε, και ως Επιτροπή δική μας και μαζί με την Επιτροπή Περιβάλλοντος ίσως. Ε, merci, Madame la Présidente.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 et évidemment une surveillance accrue en post commercialisation pour ne pas passer à côté d'effets indésirables, inattendus et qui peut έτσι, συνέχιση των ελέγχων έτσι ώστε να μην υπάρξουν παράλληλα προβλήματα. Το θέμα της εποπτείας ε, είναι πραγματικά εξαιρετικά σημαντικό στην περίπτωση των εμφυρευμάτων ε, μαστού στη Γαλλία, ε, στην υπόθεση PIP δηλαδή, οι ξαφνικές επισκέψεις και η ξαφνική έλεγχη ήταν αυτοί οι οποίοι ξεσκέπασαν το σκάνδαλο. Το ζήτημα είναι βεβαίως όσον αφορά το κείμενο ότι πρέπει και οι Κομισιόν και τα κράτη-μέλη να είναι συνυπεύθυνα. Στην διάσκεψη των Προέδρων δεν επιτύχα επιτύχαμε τη διαδικασία άρθρου 50, αλλά επιτύχαμε το 49 συν, πράγμα που μας ε, επιτρέπει ε, να ε, εκπονήσουμε γνωμοδότηση και στην ένδυ ε, γνωμοδότηση επί του συνόλου και δεν υπάρχει επομένως καταμερισμός άρθρο ε, θα γίνει μια γνωμοδότηση επί του συνόλου. Ε, η δε διαδικασία άρθρου 49 συν μας δίνει τη δυνατότητα να ξεπεράσουμε την απλή διαδικασία και επομένως να μπούμε σε συζήτηση στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου. Αυτά ήθελα να σας πω. Ε, βεβαίως θα έχουμε τη δυνατότητα να επανέλθουμε, να ξανασυζητήσουμε και αν το επιθυμείτε κυρία Πρόεδρε και αν ε, αυτή είναι η επιθυμία των ε, περισσότερων μελών της Επιτροπής βεβαίως μπορούμε να οργανώσουμε ακρόαση έτσι ώστε να έχουμε επιπλέον ε, πληροφορίες για αυτό το πολύ τεχνικό και ιδιαίτερο απαιτητικό κείμενο. Ευχαριστώ κυρία Μπέρα. Τώρα το χρονοδιάγραμμα. σχέδιο γνωμοδότησης 3 Απριλίου θα μεταφραστεί, 25 Απριλίου θα συζητήσουμε διεξοδικά εδώ στην Επιτροπή και πάλι. Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι η 6η Μαΐου, έχετε χρόνο. Και μετά η εξέταση 29 Μαΐου και οι συμβιβαστικές θα συζητηθούν στις 12 Ιουνίου. Η ψηφοφορία θα γίνει στις 18 Ιουνίου. Έχουμε χρόνο πολύ. Όλα τα άλλα θα τα συζητήσουν οι σκιώδεις. Τώρα λύεται η συνεδρίαση η επίσημη δημόσια.